τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Καλημέρα σε όλους τους αξιότιμους συναδέλφους, άντρες και γυναίκες. Ξεκινάμε τη συζήτησή μας. Ξεκινά η συνέδριαση. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά την σύσταση της κυρία Σοφή Ιντβέλτ όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών ε, στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Τώρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την συνάδελφο κυρία Σοφία Ιντβέλτ, για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον κύριο Επίτροπο. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, αυτή η διαδρομή που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003 και για αυτόν τον λόγο έχουμε και αυτήν την υπερατλαντική συμφωνία όσον αφορά την κοινοποίηση των δεδομένων ε, η διαδρομή εννέα ετής και ήδη μπορούμε να εξαγάγουμε ένα συμπέρασμα. Ε, αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί στη σκέψη ότι είναι πάρα πολύ θετικό μετά από εννέα χρόνια με τον πιο στενό μας ε, ε, σύμμαχο και φίλο καταλήγουμε σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο και σε μια, μια συμφωνία η οποία μόνο κατά το ίμιση μπορούμε ότι είναι ικανοποιητική. Είναι επομένως αυτό πάρα πολύ θλιβερό για να δούμε ποια είναι η σχέση μας με τους, ε, αυτούς τους στενούς συμμάχους και γιατί εμείς να, έχουμε τέτοια στάση ως προς εκείνους. Στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών πριν από λίγες εβδομάδες ψήφισε δυστυχώς αρνητικά για τη δική μου σύσταση ε, να καταψηφίσουμε. Και επομένως η θέση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών είναι ε, το ότι θα πρέπει να εγκριθεί η ε, συμφωνία. Και είναι για μένα θλιβερό το ότι όλοι, όλοι, ακόμα και εκείνοι που θα ψηφίσουν σήμερα ναι, όλοι ακόμα έχουν κάποια ερωτήματα. Πάντως, πρώτα-πρώτα θα ήθελα κάτι να σας πω για ένα νέο στοιχείο, δηλαδή την δήλωση της Επιτροπής, την οποία λάβαμε χθε και πραγματικά για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Δεν περιέχει νέα στοιχεία. Απλώς πρόκειται για την ε, ε, ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δεσμεύει τη είπα ούτε για εμά μας αλλάζει επομένω ε, την γνώμη. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση Γκουέ να υποβληθεί ε, το κείμενο η το Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο, δεν καταλαβαίνω, είναι συμπαθη η πρόταση και δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αναλάβουμε εμεί ω κοινοβούλιο τι ευθύνε μα. Έχουμε επίσης και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να θέσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τη δική της ερμηνεία ε, για το άρθρο 4 όσον αφορά ε, τον περιορισμό για τον σκοπό. Πάντως, θα θέλαμε πολλοί από εμάς εδώ να μάθουμε για το πώς καταλήξατε στο ότι η συστηματική χρήση των δεδομένων για άλλους στόχους ε, ρητός να εξαιρείται. Δεν καταλαβαίνω ποια διατύπωση, ποιε λέξει του άρθρου 4 σα οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Πώ συμπεραίνεται ότι η χρήση των δεδομένων για μετανάστευση, για υγεία, για τελωνία, πώς αυτό ε, αποκλείει τη χρήση των δεδομένων και πώς ε, αυτό απορρέει από τα άρθρα 82 και 87 όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία. Είπαμε πολλά όσον αφορά την περίοδο της ε, κράτησης των στοιχείων, και παρακαλώ να μου... Ε, ε, είπατε για το push και pull ότι ε, μόνο σε συγκεκριμένε περιπτώσει τα χρησιμοποιείτε αλλά γι' αυτό και θέλω να μα πείτε τι γίνεται όσον αφορά κάποιες αεροπορικέ εταιρείε ευρωπαϊκές για το 2010 και το 2011 έχουμε εδώ κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι αυτή η χρήση του pull ad hoc γίνεται δεκάδες χιλιάδες φορές ανά ημέρα. Έχουμε εδώ πέρα ε, ένα στοιχείο που μας που λέει ότι σε κάποιες συγκεκριμένες μέρες είχαμε 82.500 χρήσεις τέτοιες, τέτοιο, αυτό το πουλ. Um, the agreement explicitly says that um, uh, no rights can be derived from this agreement. Οπότε αυτό, αυτά απορρέουν από, το, από τη, τη συμφωνία αυτή. Yeah. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε τι χρήση θα γίνεται ε, από πλευρά και άλλων νομικών προσώπων. Να δούμε επίση και τι είδου δυνατότητα υπάρχει προσφυγή στη δικαιοσύνη από πλευρά των Ευρωπαίων. Τώρα ξέρω ότι τελείωσα όμω προ την ε, διάθεσή μου και θα χρησιμοποιήσω τον υπόλοιπο που έχω να δευτερολογήσω. Ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ κυρία Εντεβέλτ. Μποζόκοφ, επόμενος αγωγητή εν του Συμβουλίου. Ο κύριος Μποζόκοφ. Ευχαριστώ. Λέει ο του Συμβουλίου. Αξιότιμα μέλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Μάστρο, ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να σας μιλήσω επί τη ευκαιρία της συζητήσεως του σημαντικού αυτού ζητήματος και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγματι. Θα ήθελα να εστιαστώ επί κάποιων γενικών πτυχών που θεωρώ ότι δημιουργεί αυτό το σχέδιο συμφωνίας. Οι πιο τεχνικέ πτυχέ ε, της μπορούν να μείνουν ε, για ανάλυση στην κυρία Μάστρομ για την ώρα. Μπα τα εξηγήσει. Το θέμα λοιπόν της ανταλλαγής πληροφοριών επιβατών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεω και ΕΠΑ ΕΕ, ε, επί σειρά ετών ήταν στα, στο πρόγραμμα του Διατλαντικού Διαλόγου. Ταυτόχρονα Έχουμε λάβει ε, κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τη σημασία που έχει χρήση των πληροφοριών PNR, αλλά μόνο από τη μία πλευρά. Ε, βασικό επιχείρημα είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του συνοριακού εγκλήματος. Κατά την άποψή μου, αναμφισβήτητα, οι πληροφορίε επιβατών PNR είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την επιβολή του νόμου, για τις αρχές επιβολής του νόμου, στην προσπάθειά τους να πολεμήσουν τη σοβαρή εγκληματικότητα. Έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα αυτού. Αυτό ε, δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε ε, να έχουμε και κάποιες απαιτήσει, κάποιους όρους για τη χρήση των πληροφοριών αυτών από πλευρά των αρχών. Πρέπει να προστατευτεί η ιδιωτική ζωή των πολιτών μας. Και αυτό θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα όταν συζητούμε την καταπολέμηση και πρόληψη της σοβαρής ε, εγκληματικότητας. Και αυτό βέβαια ισχύει είτε μιλάμε για αρχές εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως είτε στις τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά για όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό σχέδιο συμφωνίας εμπεριέχει ε, σειρά νέων βελτιωμένων εγγυήσεων, εγγυήσεων ότι που δεσμεύτηκαν να αναλάβουν οι Αμερικανικές αρχές και πάντα εφαρμόζουν όταν επεξεργάζονται τις, αρχές, τις ε, πληροφορίες PNR. δεν είναι 100% τέλεια συμφωνία. Οι Αμερικανικές αρχές όμως προσπάθησαν αρκετά να καλύψουν τις ανησυχίες μας και τα συμφέροντά μας σε διάφορους σημαντικούς τομείς. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι η καλύτερη δυνατή υπό τις παρούσες περιστάσεις. Ε, πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι η συμφωνία που συζητούμε σήμερα δεν είναι το τέλος ε, του διατλαντικού διαλόγου όσον αφορά την χρήση πληροφοριών επιβατών PNR. Θα ήθελα να κλείσω ε, εκφράζοντας την αναγνώρισή μου διότι είδα ότι επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν έτοιμο να προασπίσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Ελάχιστες περιπτώσεις δείχνουν τόσο ξεκάθαρα όπως αυτή αυτό το μέλημα. Και θα το δείτε και αυτό να αντικατοπτρίσει τη συμφωνία που θα ψηφιστεί. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το βελτιωμένο κείμενο που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι αποτέλεσμα των επιθυμιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να Γι' αυτό σας ενθαρρύνω να υποστηρίξετε αυτή τη συμφωνία. Ε, σημαίνει ότι Εξασφαλίζουμε έτσι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι αεροπορικές εταιρείες προστατεύονται καλύτερα και στέλνουμε ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα ότι μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Αβώνας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει και να καταλήξει σε κάποια απτά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συνεργάζονται στενά όταν αντιμετωπίζουν δύσκολα καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου και τώρα το δώρο το δίνω στην κυρία Επίτροπο Σετσίλια Μάλστρομ και για σας τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργέ, η Κομισιόν συστήνει στο Κοινοβούλιο να συνενέσει για τρει λόγους τη συμφωνία. Πρώτον, και όπως εξήγησε ο Υπουργός, οι διοκτικές αρχές χρειάζονται τα PNR για να αντιμετωπίσουν τις απειλές ασφαλείας των ΗΠΑ. Δεύτερον, η συμφωνία είναι μείζον βελτίωση σε σχέση με την υφιστάμενη που ισχύει τώρα και μου μας ζητήσατε να επαναδιαπραγματευτώ. Τρίτον, είναι δύσκολο να δούμε εναλλακτικέ που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Η ανάγκη για δεδομένα PNR, η Κομισιόν έδωσε πολλές φορές στοιχεία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που δείχνει ότι τα δεδομένα PNR είναι σημαντικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της καταπολέμησης της εμπορίας ναρκωτικών και προσώπων έπαιξαν σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπίσουμε τον David Headley, τον Μοβιστή, ε, το Λονδίνο και το Μετρό, το βομβιστή στην ε, Times Square στη Νέα Υόρκη. Βοήθησαν τα δεδομένα PNR στην εξυχνίαση. Δεύτερον, Υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία του 2007. Είναι πολύ σημαντικό σε σχέση, είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το σχέδιο του Μαΐου όπου ζητήθηκε η Συμβουλή του Κοινοβουλίου και έγινε πολύ καλή συλλογική εργασία για να κάνουν οι ΙΠΑ περισσότερε παραχωρήσει. Ένα παράδειγμα πώ λειτουργεί η συνθήκη τη Λισαβόνα. Τρία θεσμικά όργανα που συνεργάζονται με σαφή μηνύματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τόσο ώστε η Κομισιόν να είναι σαφέστατη στις διαπραγματεύσεις της με τους Αμερικανούς. Το καλό συλλογικό αυτό έργο έδωσε με περισσότερη σαφήνεια, καλύτερη αμοιβαιότητα, καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών σε σχέση με την ιδιωτική, τα ιδιωτικά δεδομένα, χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των δεδομένων και η ασφάλεια ένθεν και εκείθεν του Ατλαντικού. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες σας που εκφράστηκαν στο ψήφισμα πριν από δύο χρόνια το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την αρχή της αναλογικότητας. Μπαίνω σε κάποιες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή σε σχέση με την υφιστάμενη είναι ένα ενιαίο νομικά δεσμευτικό κείμενο με γλώσσα συνθήκης. Ενισχύει την αμοιβαιότητα και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεώνοντας τη ΣΥΠΑ να, να μοιράζονται δεδομένα ε, με τις διοκτικέ αρχές και ε, στοιχεία με τις διοκτικές αρχές. Ε, είναι πιο συγκεκριμένη η χρήση των ε, PNR δεδομένων. Ε, ξέρω εδώ και τις αντιρρήσεις σας και τις αντιρρήσεις της εισηγήτριας. Θέλω λοιπόν να διαβάσω τη δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η συμφωνία ε, θεσπίζει συγκεκριμένη περιγραφή πεδίου εφαρμογής ε, διευκρινίζοντας το σκοπό για τη συλλογή και χρήση των στοιχείων PNR. Υπάρχει λεπτομερής ε, αναφορά στο σκοπό των στοιχείων στο άρθρο 4 που συνάδει με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική σφαίρα. Είναι, περιορίζονται στην πρόληψη, ανείχνευση, ανάκριση, δίωξη, τρομοκρατία δημοκρατικών αδικημάτων και διακρατικών ε, εγκλημάτων. Ε, για πρώτη φορά ορίζονται τα τρομοκρατικά αδικήματα και τα διακρατικά εγκλήματα. Στο 4.1, στο 4.2 υπάρχει η δυνητική χρήση των PNR δεδομένων σε βάση ad hoc για την προστασία ζωτικών συμφερόντων ή ουδήποτε ατόμου ή αν ζητηθεί από δικαστήριο. Αυτές οι χρήσεις εκφύσεως και με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε από, τις κοινές, από τους κοινούς ελέγχους είναι η εξαίρεση. Στο 4.3 διευκρινίζεται πώς τα PNR είναι σημαντικά όταν ε, ταξιδεύουν από ή προ τις η οι επιβάτε. Διευκρινίζεται ότι τα PNR σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογή του σκοπό του, μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εξέταση το 4-4 εξηγεί ότι η συμφωνία δεν προδικάζει το, την εθνική νομοθεσία, τις εθνικές αρμοδιότητες ε, ε, όταν ε, εντοπίζονται ε, ε, προβλήματα στη χρήση των στοιχείων PNR η διευκρίνηση ε, αυτή δεν επεκτείνει την χρήση δεδομένων PNR. Στα πλαίσια του κοινού μηχανισμού αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 22 και χωρίς να προδικάζονται άλλα θέματα που μπορεί να τεθούν στα πλαίσια του μηχανισμού, η Κομισιόν ζητεί συγκεκριμένες πληροφορίες λεπτομερείς σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 4. Πιο συγκεκριμένα θα επανεξετάσει τη χρήση των στοιχείων PNR ε, βάσει του άρθρου 4.1 θα ζητήσει πληροφορίε για οποιασδήποτε περιπτώσει όπου τα PNR χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία ζωτικών συμφερόντων και όπου ζητήθηκαν ε, από το δικαστήριο βάσει του άρθρου 4.2 τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεσμεύεται να ενημερώνει πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα τα θέματα ε, και να υποβάλει πλήρη έκθεση στο Κοινοβούλιο όπω προβλέπει το άρθρο 23.3 αμελητή στο τέλος της, πρώτης, της του πρώτου κοινού ελέγχου. Ε, μετά τον κοινό έλεγχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα εκφράζει την απόψη, τις απόψεις του σε σχέση με τις ελλείψεις και καλεί την αναστολή η πάυση της συμφωνίας. Η Κομισιόν ε, δεσμεύεται να εξετάζει το πολιτικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη μέγιστη προσοχή για να αποφασίσει αν θα υποβάλει πρόταση ε, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 218 της συνθήκης. Πάμε τώρα σε άλλα σημεία μετά το πεδίο εφαρμογή. Η συμφωνία ε, μειώνει την περίοδο φύλαξη δεδομένων ε, από 15 σε 10 χρόνια για σοβαρά διακρατικά εγκλήματα. Μόνο για τρομοκρατικά αδικήματα τα δεδομένα θα φυλάσσονται για 15 χρόνια όπω ε, είναι στην τωρινή συμφωνία. Και ένα καινούριο σημαντικό στοιχείο. Ε, θα ανωνυμοποιούνται τα στοιχεία PNR έξι μήνες αφότου στέλνονται και αυτά δεν θα μπορούν πια να οδηγήσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διατάξεις για την προστασία δεδομένων, ειδικότερα για τον παράνομο προσδιορισμό χαρακτηριστικών, το profiling. Ε, είναι πολύ σημαντικό κάποιος άνθρωπος να λαμβάνει την τελική απόφαση ε, και όχι οι διαδικασίες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χάνονται ή να αποκαλύπτονται στα δεδομένα. Επίσης ε, προσδιορίζονται ε, τα, οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση αλλά και για τη διαγραφή των δεδομένων. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες ε, διατάξεις με βάση το Αμερικανικό Δίκαιο. Επίσης ε, μπορούν ε, δεδομένα να χρησιμοποιούνται ε, όχι συλλογικά αλλά σε ατομική βάση για συγκεκριμένες χρήσεις. Είναι πολύ σημαντική η συμφωνία σχετικά με τη διαβίβαση. Η μέθοδος είναι η μέθοδος push μέσα σε δύο χρόνια δεσμεύθηκε η Κομισιόν ότι μπορεί να γίνει αυτό από τις αεροπορικές εταιρείε. Στοιχεία πουλ δεν θα απογορεύονται τελείως, αλλά οι συνθήκες περιορίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην τωρινή συμφωνία ε, η μέθοδος πουλ δεν είναι ο κανόνας. Τώρα γίνεται ο κανόνας, ενώ η μέθοδος πουλ είναι κατ' και θα ελέγχεται καθ' ολοκληρία από την Κομισιόν όταν εφαρμόζεται. Τέλο, υπάρχουν διατάξει που διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται σωστά η συμφωνία υπάρχουν ανεξάρτητοι έλεγχοι από διάφορους φορείς ε, μέσα και έξω από το Υπουργείο Εσωτερική Ασφάλεια. Θα γίνεται πλήρη αξιολόγηση μετά από τέσσερα χρόνια. Θα υπάρχουν ε, αρχεία, logs, ε, υπάρχουν επίσης διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ ημών και των ΙΠΑ και διαδικασίες που προβλέπουν την αναστολή ή την πάυση. Ε, η απόφαση είναι ε, δύσκολη σχετικά με τη συμφωνία. Είμαι διατεθειμένη να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Η διεθνή συμφωνία. Δεν είναι 100%. Είναι διεθνής η συμφωνία, όπως όλες οι διεθνείς συμφωνίες δεν είναι 100% τέλεια. Πρέπει να υπάρχει δούνε και λαβήν. Η Κομισιόν παρουσίασε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ένα σχέδιο συμφωνίας του Μαΐου. Εκεί δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για το τι αλλαγές θα γίνουν πήγαμε πίσω και επιτύχαμε με τη ΣΥΠΑ πολλέ από τι αλλαγέ. Για τον περιορισμό του σκοπού, για το πεδίο εφαρμογή, για την περίοδο φύλαξη των δεδομένων και άλλα στοιχεία. Και έχουμε τώρα μια συμφωνία που σέβεται απόλυτα το δίκαιο το δικό μα. Και περνώ στο τελευταίο θέμα. Ε, έλλειψη καλύτερων εναλλακτικών περαιτέρω διαπραγματεύσει, με τη ΣΥΠΑ δεν αποτελούν πραγματική επιλογή. Τι θα γίνει λοιπόν αν απορρίψετε σήμερα τη συμφωνία. Αυτό θα είναι επιζήμιο για τις διατλαντικές σχέσεις, διότι τα δεδομένα αυτά θα συλλέγονται ούτως ή άλλως και θα χάσουμε πολύ σημαντικές ε, δυνατότητες να επηρεάσουμε την αμερικανική πολιτική για τη χρήση αυτών των δεδομένων. Δεύτερον, οι αεροπορικές εταιρείε θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση, διότι θα τους ζητηθεί να διαβιβάζουν τα δεδομένα, αλλά δεν θα υπάρχει νομική βάση στην, νομική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διαβιβάσεις των δεδομένων. Αυτό λοιπόν θα μας δημιουργήσει νομικό κενό, νομική αφάνεια και θα υπάρχει πρόβλημα για τους επιβάτες και πολύ δύσκολη κατάσταση. Τέλος, πολύ σημαντικό, δεν θα μπορέσουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των άνω των 48 εκατομμυρίων επιβατών που πηγαίνουν στη ΣΥΠΑ κάθε χρόνο. Ελήψη συμφωνίας δεν θα υπάρχει δεσμευτικός διεθνής κανόνας για να προστατευτεί η ιδιωτική σφαίρα των επιβατών. Μπορεί βέβαια να υπάρξουν διμερείς συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και τα κράτη-μέλη μας, αλλά δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη διμερώς θα μπορέσουν να επιτύχουν προστασία επιβατών μεγαλύτερη από αυτή που επιτύχαμε σήμερα. Για όλους αυτούς τους λόγους σας ζητώ σήμερα να εγκρίνετε την ε, συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μάστρο. Ουγγουρεάνου το επόμενο όνομα. Μπράιαν Ουγγουρεάνου για δύο λεπτά. Απουσιάζει και ο Καλώς. Εν ονόμα των κοινοβουλευτικών ομάδων οι αγορητέ. Πρώτο όνομα Βο, για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την ε, εξαιρετική και υποδειγματική δουλειά. Πολύ από την κριτική της Σόφη Ίνφελτ με βρίσκει σύμφωνο και εν μέρη την ε, υποστήριξα. Όμως ε, υπάρχει ένα σημείο στο, όπου πρέπει κανείς να αναλάβει τις ευθύνες του. Για το ΕΛΚ και προσωπικά πρέπει να πω ότι τώρα πρέπει να μας απασχολήσει η πραγματικότητα και όχι η ιδεολογία ή θεωρητικά επιχειρήματα. Γεγονός είναι ότι είπα εδώ και 10 χρόνια συλλέγουν δεδομένα PNR και δεν υπήρξε ούτε μία προσφυγή. Ε, η καταγγελία. Βεβαίως και δεν θέλουμε η ε, διαβίβαση δεδομένων να σταματήσει. Αυτό το είπατε κι εσείς. Γεγονός επίσης παραμένει ότι δεν θέλουμε οι αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ να σταματήσουν. Γεγονός επίσης είναι ότι οι ΙΠΑ έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος ε, ε, εισέρχεται στη χώρα τους. Γεγονός είναι θεωρώ ότι οι νομικές υπηρεσίες ε, μας είπαν όλες ότι αυτή η συμφωνία είναι καλύτερη από την προηγούμενη συμφωνία και τις εναλλακτικέ. Άρα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε εκλεγεί. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για τους πολίτες που κατά τα άλλα θα αφήναμε με λιγότερη προστασία. Ευθύνη απέναντι στις αεροπορικές εταιρείες και το επίσης αυτό η Επίτροπος που θα βρίσκονται σε ανασφάλεια δικαίου. Πρέπει να αναλάβουμε επίσης και ευθύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, διαπραγματευτικό εταίρο σε θέματα ασφάλειας ε, να αναλάβουμε ευθύνη για ισορροπημένη σχέση μεταξύ ασφάλειας από τη μία πλευρά και προστασίας δεδομένων από την άλλη. Γι' αυτό, σούμα ε, έστω εν γνώση ότι δεν είναι τέλεια η συμφωνία, κρίνοντας όμως τις συνέπειες ε, που θα είχε η μη συμφωνία, ε, επιλέγουμε να την εγκρίνουμε και έτσι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Προτείνω λοιπόν την υπερψήφιση της συμφωνίας. Κύριε Βος, δέχεστε να σε υποβληθεί μια ερώτηση εκ μέρους της κυρίας Ιντβέλτ. Σας παρακαλώ, κύριε Ιντβελτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση να απευθύνω προς τον κύριο Βος και την πολιτική τομάδα. Σωστά είπατε ότι πρέπει να υπάρχει νομική βάση για τη μεταφορά στοιχείων επιβατών. Διρωτώ λοιπόν γιατί το Κοινοβούλιο δεν αντέδρασε στο γεγονός για το οποίο επί 3,5 χρόνια στοιχεία δόθηκαν στον Καναδά αντί απουσία εσδήποτε νομικής βάσεως και με το πρόγραμμα ασφαλών τρίσεων τον είπα, μεταφέρονται στοιχεία από την Ευρώπη προ τι Ηνωμένε Πολιτείε για πτήσει που δεν πηγαίνουν στι Ηνωμένε και το Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να νοιάζεται. Γιατί θέλουμε νομική βάση σε μία περίπτωση και όχι στην άλλη. Ορίστε, απαντήστε. Ευχαριστώ. Καταρχήν πάντα θέλουμε νομική βάση και τώρα είναι ατυχής η κατάσταση με τον Καναδά. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Από την άλλη, τα δικαιώματα υπερπτήσεων ε, αφορούν και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλου κράτους. Χρειάζονται λοιπόν και εδώ ε, σαφείς βάσεις. Πρέπει να υπάρχει βάση. Αν λείπει χρειάζεται να ε, προσθεθεί και δεν είμαστε κατά της νομικής βάσης εν προκειμένου, απλώς περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τον Καναδά. Αυτά περιμένουμε. Και βεβαίως θα ε, ζητήσουμε να συμπεριλαμβάνεται και στη συμφωνία εκείνη νομική βάση. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Κλοντ Μωράες έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ από σοσιαλιστών και δημοκρατών, εμείς θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Και είχαμε μια ελαφρά πλειοψηφία υπέρ στην Επιτροπή. Όπως τα ακούσατε ε, από διάφορους και τους σκιώδες. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ από δύο εξή Είχαμε εμείς τρεις βασικούς στόχου. Θεωρήσαμε ότι αυτή η συμφωνία ε, φυσικά ε, επειδή έχετε βελτίωση αλλά από την άλλη μεριά ότι καλύπτει πάρα πολλούς στόχους του της τρομοκρατίας μεγάλη περίοδο κατακράτησης ε, των στοιχείων δύο από τις τρεις παραχωρήσεις είπαμε ότι είναι αρκετό ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η η κρίση μας διαμορφώθηκε έτσι θετικά. Ήταν πάντως δύσκολο να διαμορφώσουμε αυτό το συμπέρασμα. Τώρα όμως έχουν βγει κάποια εγκλήματα, κατακράτηση επίσης μειώθηκε και ξέρουμε ότι είπα δεν θέλουν να υποχωρήσουν σε όλο το push και pull. Ε, τώρα θα υπάρξει χρήση σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια σοβαρή, μεγάλη απειλή και ιδίω για το push and pull ε, δεν ικανοποιηθήκαμε αλλά θα πρέπει κάπου να καταλήξουν αυτές οι τόσο πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις και κατά τη γνώμη μια ελαφρά πλειοψηφία συμφώνησε ότι οπωσδήποτε έχουμε βελτίωση του κειμένου και έτσι θα έχουμε την διαδόση των δεδομένων και όπως είπαν πολλοί έτσι διαμορφώνουμε μία συμφωνία και έτσι δεν θα έχουμε 27 χωριστές διμερείς. Δεν θα υπάρχει νομικό κενό. Δεν θα έχουμε αντιφάσεις στην ε, ρύθμιση της υπόθεσης, για το οποίο δεν εξυπηρετεί κανέναν. Όσον αφορά τώρα το προηγούμενο που δημιουργείται, δεν θεωρούμε ότι ισχύει κάτι. Δεν υπάρχει ούτε από τη μία ούτε συμφωνία προηγούμενα. Συνολικά η κατάσταση είναι ικανοποιητική, δεν είναι ιδανική, τέλεια, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάνει τη να λάβει υπόψη σοβαρά το Κοινοβούλιο. Επίτροπε, εμείς τώρα βοηθούμε και εσείς να λάβετε υπόψη τη δική μας γνώμη και να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, αν τα πράγματα ξεφύγουν πέρα από την εντολή σας. Ευχαριστώ. Ρενάτε Βέμπερ για δύο λεπτά. Κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι επίμαχη η συμφωνία αυτή. Ο στόχος μένει πρόσδεκτος η καταπολέμηση τρομοκρατίας μέσω προληπτικών μέσων. Όμως, δε, παρεμβάλλεται στην προστασία της ιδιωτική ζωής και την προστασία των στοιχείων. Αυτό είναι διαφυσβήτητο. Δεν είμαι η μόνη που λέγει ότι η συμφωνία παραβιάζει τα λόγω δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων το παρουσίασε αυτό διεξοδικά σε μια ανάλυση. Και το πεδίο διεφαρμογής της ε, εφαρμογής ξεπερνά τα όρια της καταπολέμησης απλώς της τρομοκρατίας. Μερικοί θεωρούν ότι αυτή είναι καλύτερη συμφωνία από την προηγουμένη. Αυτό σημαίνει μόνο ότι είναι λιγότερο κακή από την προηγουμένη. Όμως παραμένει μια συμφωνία που έχει σοβαρέ συνέπειε όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά μα. Σέβομαι το ότι οι Αμερικανικέ αρχέ και οι νομοθέτες ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των πολιτών τους. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα να νοιαζόμαστε πάνω απ' όλα για την προστασία των δικών μας Ευρωπαίων πολιτών και των δικαιωμάτων τους. Έχει υποθεί ότι χωρί τη συμφωνία οι αεροπορικέ εταιρείε μα θα παραβιάσουν την νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση την προστασία των δεδομένων, διότι αν θέλουν να προσγειωθούν στι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διαβιβάζουν στοιχεία αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η συμφωνία υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείε να εφαρμόσουν την υποχρέωση που ε, σε δύο χρόνια να στέλνουν τις πληροφορίες, άρα πρέπει να ξοδέσουν πάρα πολλά χρήματα σε εξοπλισμό και λογισμικό για να διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία στις ΗΠΑ σε πραγματικό χρόνο. Τι γίνεται αν κάποιες αεροπορικές εταιρείε δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις υποχρεώσεις. Μεγάλες εταιρείε πιθανότατα θα τα καταφέρουν, αλλά μικρότερες εταιρείε είτε θα χρεοκοπήσουν λόγω αυτών των δαπανών, είτε η παρούσα κατάσταση θα συνεχιστεί. Θα επιτρέπουν την άντληση πληροφοριών πλευρά Αμερικανικών αρχών που θα παίρνουν τα στοιχεία από του δικού υπολογιστέ. Ποτέ δεν πίστεψα ότι ένα κακό νόμο είναι καλύτερο από καθ... να μην υπάρχει νόμο. Ευχαριστώ, κυρία Βέμπερ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα για δυόμιση λεπτά, Άλμπρεχτ, ο κύριο Άλμπρεχτ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, πριν από περίπου τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, εξέδωσε σημαντική απόφαση σε σχέση με τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Διαπιστώνει ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων σε κεντρικές βάσεις δεδομένων των κρατών ε, αντιβαίνει στον νόμο, στο δίκαιο. Πριν από δύο χρόνια το Γερμανικό Ομοσπονδιακό δικαστήριο ε, ε, αποφάσισε σε σχέση με τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και αποφάσισε ότι ακόμα και για λίγους μήνες ε, η φύλαξη δεδομένων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παρόλα αυτά ε, καλούμεθα να δεχθούμε μια συμφωνία που ούτε κατά προσέγγιση δεν ε, συνάδει με τις ε, αποφάσεις των δικαστηρίων. Φύλαξη δεδομένων μέχρι 15 χρόνια είναι δυσανάλογο μεγάλο διάστημα. Είπαμε ότι ο σκοπός φύλαξης αυτών των ε, δεδομένων μπορεί να ισχύει για δεδομένα που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Επίση, ο προσδιορισμό δεδομένων profiling των πληροφοριών δεν επιτρέπεται. Επίση, αγαπητή κυρία Μάλφρεμ, σε αυτή τη συμφωνία με αυτά τα μέτρα όλα τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται και θα την χάνουν επεξεργασία. Δεν ε, θα χρησιμοποιούνται ε, συγκεκριμένα δεδομένα, αλλά όλα. Ε, είναι λοιπόν αυτή μία ε, διαδικασία αυτοματοποιημένη η οποία ε, ε, περιλαμβάνει το profiling. Ε, είναι λοιπόν αυτό ανοιχτή σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδιαίτερα θα ήθελα να πω προς τους συντηρητικούς και τους σοσιαλδημοκράτες θα ήθελα να ρωτήσω δεν τρέπεστε τόσο κατάφορα να παραβιάζετε το δίκαιο στο Κογκρέσο των είπα η τα μέλη του Κογκρέσου θα έδιναν πιο ε, αποφασιστική μάχη για τα δικαιώματά τους. Εμείς ε, θα νομιμοποιήσουμε τέτοιες πρακτικές ως Ευρωπαίοι. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τέτοιες πρακτικές. Ε, πολλοί πολίτες είναι απογοητευμένοι και θα απογοητευτούν ακόμη περισσότερο αν μετά από 10 χρόνια αντιπαράθεσης το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή τη συμφωνία που ακόμη περιλαμβάνει όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό ε, τιμήστε το κύριο του Κοινοβουλίου και ψηφίστε κατά. Κύριε Άλμπρεχτ, κύριο Μορβάη θα ήθελα να σε απευθύνει ε, ένα ερώτημα. Δεχόσαστε. Κύριε Άλμπρεχτ, συμφωνείτε να δεχτείτε ερώτημα. Ναι, ορίστε. κυρία Μορβαέ, Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο της. Α, λειτουργεί τώρα. Μία ερώτηση προς διευκρίνηση. Συμφωνώ σχεδόν απόλυτα μαζί σας, κυρίω λαμβάνοντα υπόψη τι τεράστιε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξε η κυβέρνηση την οποία συζητούμε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Θέλω διευκρίνηση επί του θέματος της αναλογικότητας σε σχέση με το σκοπό, διότι για πολλούς κυρίως τους μη νομικούς, ίσως να είναι ανησυχητικό αυτό. Διότι παρετούμενοι από κάποια στοιχεία, από κάποια δικαιώματα προστασία ιδιωτική ζωής ίσως αυτό να είναι ανάλογο με τον αξιέπαινο στόχο της πρόληψη ε, της τρομοκρατίας Ε, αυτού συμφωνούμε όλοι, πιστεύω. Το ερώτημα είναι, αυτός ο αξιέπαινος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί πράγματι μέσω των μέτρων που λαμβάνονται εδώ. Και εδώ έχω πρόβλημα εγώ και γι' αυτό θα ψηφίσω όχι σήμερα. Και ποια είναι η άποψή σα επ' αυτού. Αναλογικότητα έναντι στόχου, έναντι σκοπού. Ε, διευκρίνηση επ' αυτού. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ του συναδέλφου να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο ε, τη γαλάζια κάρτα. Κύριε Άλμπρεχτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την διευκρινιστική ερώτηση. Βεβαίω η καταπολέμηση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματο είναι απαραίτητο στόχο, και θεωρώ ότι είναι σημαντικό μέτρο ε, που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους συμμάχους μας τη είπα ε, Αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά μπορούμε να πετύχουμε το στόχο με τη μαζική ανάλυση δεδομένων πολλών ανθρώπων που δεν θεωρούνται ύποπτοι, δεν είναι ύποπτοι ή χρειάζεται περισσότερο μια ενισχυμένη συνεργασία όταν υπάρχουν υποψίες ε, ε, συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών, αστυνομικών αρχών. Εκεί θα πρέπει να, προς εκεί θα πρέπει να πάμε. Δίνουμε πολλά χρήματα για ε, κέντρα δεδομένων, κέντρα αναλύσεων, όπου αναλύονται δεδομένα μη υπόπτων, ενώ από την άλλη πλευρά... δεν επικεντρωνόμεθα στην στο αστυνομικό έργο με τους υπόπτους. Πηγαίνουμε τώρα ε, στον κύριο Κίρκοπ για δύο λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το τι κάνουμε εδώ χαρακτήρισαν πάρα πολύ διφορούμενη αυτή τη συμφωνία, αλλά οι βελτιώσει κατόπιν όλων των διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ήταν κάτι το οποίο βρήκε τη συνένεση των πέντε παρατάξεων του Συμβουλίου και τη Κομισιόν. Εγώ διαφωνώ με την εισηγήτρια γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι σχετικέ βελτιώσεις ε, παρά βέβαια αυτό πάρα πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διαπραγματεύση μεταξύ των δύο πλευρών πρόεδρε του ε, οποιονδήποτε δύο οποιασδήποτε διαπραγματεύσει ποτέ θα οδηγήσουν σε κάτι το οποίο είναι τέλειο, ιδανικό. Αυτό δεν θα πρέπει κανεί να το προσδοκά και να το παραμείνει. Όμω, όμως, είναι ο πιο έμπιστο εταίρο μα. Ε, είπα και ότι αυτά τα οποία έγιναν στην πρόσφατη ιστορία δεν θα πρέπει κανεί να τα ξεχνά και να τα αγνοεί. Ούτε επίσης ε, θα πρέπει να ξεχνούμε το πόσο ε, έχει, έχει, έχει, έχει δικαιωθεί η χρήση αυτών των ε, δεδομένων PNR κατά εγκληματιών και τρομοκρατών σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξή. Τι αναλυτική λύση υπάρχει, 27 διμερείς συμφωνίες. Έτσι θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου, θα υπάρχει σαφές νομικό δεν θα έχουν ε, προσβασιμότητα στην δικαιοσύνη οι επιβάτες. Όχι, δεν υπάρχουν εναλλακτικέ παραδεκτές από το Κοινοβούλιο. Και όσοι εδώ δεν θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι κάτι το αναγκαίο, ας εξηγήσουν τους λόγους στους ψηφοφόρους. Όχι πολιτικά μας μάθα ψηφίσουμε υπέρ, γιατί ξέρουμε ότι τελικά αυτή η συμφωνία δεν είναι η τέλεια. Όμως αποτελεί ένα ακόμα μέσο για εξασφάλιση ε, των Ευρωπαίων από ασφάλεια. Ακριβώ έχουμε το δικαίωμα και έχουν οι Ευρωπαίοι το δικαίωμα να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ κύριε Κερκόπ. Έχουμε δύο αιτήματα για υποβολή ερωτήσεων για σας. Κύριε Κύρκοπ, δεχόσαστε να αποδεχτείτε, δεχόσαστε τις δύο που να σας υποβάλουν. Πρώτη ερώτηση του κυρίου Βότσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να προσπαθήσω να προσπαθήσω του Ευρωπαίους κατά της δημοκρατίας και αυτό ε, είναι κοινό μεταξύ ημών και των Αμερικανών συμμάχων. Όμω θα πρέπει αυτό να γίνεται με αλληλοσεβασμό. Και θέλω τον κύριο κύριο να τον ρωτήσω το εξή επί βάση της ε, εμπειρίας του. Κύριε Κέρκοπ. Εάν κανείς ε, ρωτήσει τον Αμερικανό νομοθέτη και του πει να νομοθετήσει κατά της δικής νομοθεσίας και έτσι να, κάνει, να νομοθετήσει αντιβαίνοντας τη νομική του παράδοση. Τι λέτε, τι θα πει ο Αμερικανός νομοθέτης. Ορίστε, απαντήστε. Μου αρέσουν πολύ υποθετικές συζητήσεις, Πρόεδρε. Κυρίως όταν συζητούμε κάτι που είναι τόσο σημαντικό. Μπορώ να πω με κάποια βεβαιότητα, πιστεύω, δεν είμαι Αμερικανός, γνωρίζω πολλούς Αμερικανούς νομοθέτες, όπως και ο Σαργκρέμ, όμως έχω την πεποίθηση ότι οι νομοθέτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποφάσισαν να κάνουν ό,τι θα ήταν αναγκαίο για να προστατεύσουν όχι μόνο τους δικούς τους πολίτες, αλλά και τους άλλους πολίτες του ελεύθερου κόσμου με τους οποίους έχουν ε, συναλλαγές. Και αυτή είναι η εμπειρία μου από τη είπα. Ίσως να είναι οι ίδιες εμπειρίες για όλους, αλλά πιστεύω ότι αυτές θα ήταν οι προτεραιότητες τους. Και τώρα η κυρία Ίντβερτ θα υποβάλει ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσεις προς τον συνάδελφο Κέρκοπ. Είπατε ότι πρέπει να αποδεχθούμε το κύρος της νομικής υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την άποψή τη. Εσεί δεχόσαστε το κύριο τη ε, Εποπτική Αρχή Υποστασία των Δεδομένων και την ομάδα του άρθρου 29 που λένε και οι δύο φορεί ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί παράβαση του νόμου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεύτερο ερώτημα. Σωστά αναφερθήκατε σε θέματα ασφαλεία. Γιατί όμω οι συντηρητικοί πάντα ανησυχούσαν για εύκαμπτη κυβέρνηση, όχι μεγάλη κυβέρνηση. Γιατί θέλετε να, χρησιμοποιούνται για σκοπούς υγείας μετανάστευσης, και τελωνιακή πολιτική αυτά τα στοιχεία. Ορίστε. Απάντηση. Πρόεδρε, δεν έχω πρόθεση να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα, διότι θεωρώ ότι είναι θέμα για άλλη περίσταση. Κυρία Ιντβέλτ και εγώ κατηδίαν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Όσον αφορά του νομικού και τι απόψει, ω νομικό, εγώ με... έχω συνηθίσει να εκφράζω γνώμε. Δεν πιστεύω ότι ακολουθείται η άποψή μου σαν μονομένο νομικό απόλυτα ούτε ότι κάποια ομάδα νομικών έχει μονοπόλιο όσον αφορά την ορθότητα μιας απόφασης. Εγώ πιστεύω ότι η νομική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η βασική νομική προ του οποίου θα έπρεπε να απευθυνθούμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα αστικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα εκ μέρου μα, όσον αφορά τις διεθνείς μας συμφωνίες που συνάπτουμε. Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι η νομική άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η βασική γνωμοδότηση στην οποία θα έπρεπε να βασιστεί και βασίζομαι από αυτής. Και κατά πόσο άλλες νομοδοτήσεις ήταν εξίσου σημαντικές, αυτό είναι θέμα ε, πλαισίου εντός το οποίο για τη συζήτηση. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μπάτεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις περιορίζουν όλο και περισσότερο την ιδιωτική σφαίρα και την ελευθερία για να μας προστατεύσουν υποτίθεται από οργανωμένο έγκλημα και ε, τρομοκρατία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όμως. Δεν πρέπει να μας αφαιρεθούν οι ελευθερίες μας γιατί όταν, όταν ε, αρθούν δεν μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν. Επίσης ε, έχουμε συγκεκριμένους λόγους να εμπιστευόμαστε αυτές τις κυβερνήσεις. Ε, πρέπει η νομοθεσία να είναι ελεγχόμενη, περιορισμένη, αναλογική. Όταν θεσπιστεί η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να ε, ε, διασφαλίσουμε ότι δεν θα διευρυνθεί ανάλογα με τις κυβερνητικές επιθυμίες. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Η συμφωνία αυτή είναι διεθνής και θα πρέπει να υπογραφεί από κυρίαρχα εθνικά κράτη. Η νομοθεσία αυτή είναι απαράδεκτη όμως γιατί είναι μονόδρομος μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε για τους πολίτες μας προσωπικά στοιχεία ενώ εκείνοι δεν δίνουν τα δικά τους. Επίσης, την πρόταση ψηφίσματος θα έλει να παραπέμψει την τελική απόφαση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφανθεί σε σχέση με το αν συνάδει με την Ευρωπαϊ... το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ε, θα ψηφίσουμε κατά. Ε, δεν ε, θα ψηφίσουμε υπέρ της πρότασης ε, ψηφίσματος γιατί δεν δεχόμαστε ότι νομιμοποιείται να αποφανθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Για μισή λεπτά το λόγο έχει η κυρία Κορνίλια Ernst. Κυρίες και κύριοι, η Γκουέντζιέλ θα καταψηφίσει γιατί ένα θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών υπονομεύεται έτσι. Δηλαδή το δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ε, κυρία Μάλμστρομ, ε, μιλάτε για μια εικονική ασφάλεια που δεν διασφαλίζεται με καμία παρόμοια συμφωνία. Δεν πρόκειται για κάποια ταξιδιωτικά δεδομένα σε συνδυασμό με άλλες βάσεις δεδομένων που, υπάρχει, ε, εδώ, που υπάρχουν εδώ και καιρό. Βεβαίως και γίνεται το profiling εμείς απορρίπτουμε αυτή τη συμφωνία γιατί δεν δίνει πιστικά στοιχεία, ούτε αυτά που είπατε μας έπεισαν κυρία Μάλμστρομ, για τη χρήση αυτή της συμφωνίας. Και επειδή η αναλογικότητα και ο σκοπός ε, γίνονται παράλογες, οδηγούνται στο παράλογο όταν ε, συλλέγονται τόσα δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων. Απορρίπτουμε τη συμφωνία γιατί ξεπερνάει πολύ το πεδίο εφαρμογής που αναφέρατε. πολέμηση οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας και διασυνοριακού εγκλήματος. Ε, υπάρχει στο άρθρο 4 μια ρήτρα που πρέπει επίσης να συζητήσουμε. Μια, μια ρήτρα που ε, ανοίγει πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογής. Είναι αδύνατο να ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία γιατί η επεξεργασία των στοιχείων PNR μπορεί να δοθεί και σε τρίτες, να γίνει και από τρίτες χώρες. Μπορεί ε, ε, ε, μεταδιαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας που κοινοβουλευτικά δεν ελέγχεται. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Ε, ναι, απορρίπτουμε τη συμφωνία διότι ο χρόνος φύλαξης των δεδομένων αντιβαίνει προς οποιαδήποτε κατανόηση της αναλογικότητας και του σκοπού. Ακόμα και λογικά δεδομένα ε, που φυλάσσονται 30 μέρες αποτελούν πολλές φορές σκάνδαλο. Είναι αδύνατο να ψηφίσουμε υπέρ γιατί επίσης δεν υπάρχει και κανένα ένδικο μέσον. Ε, είναι περιορισμένο το δικαίωμα ενημέρωσης. Ε, δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, δεν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένδικα μέσα για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Θα ήθελα να πω σε όσους στάσονται υπέρ ότι εάν μας ενδιαφέρουν οι δικές μας συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν τις πιστεύουμε, πρέπει να απορρίψουμε την, απόφαση, την συμφωνία αυτή, αναλαμβάνοντας όντως ευθύνες, αλλά ευθύνες υπέρ των πολιτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Ζήλστρα είναι το επόμενο όνομα που έχω στο κατάλογό μου για μισή λεπτό. Ο κύριος Ζήλστρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. πρώτη ευθύνη των αρχών είναι η ασφάλεια των πολιτών. Και επομένω, όλοι μας οφείλουμε να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους. Έχουν δίκιο οι πολίτες να προσδοκούν την παροχή ασφάλειας. Και επομένω, γι' αυτό και πρέπει το κράτο να δημιουργήσει και τι σχετικέ εγγύσει. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν πώ να καταπολύσουν την τρομοκρατία. Όμως, η συλλογή πολλών δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουν την υποχρέωση Επομένω, καταπολέμηση τρομοκρατία από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να επομένω τι έχει γίνει ο πλευρά Αμερική, να τι έχει γίνει ο πλευρά Βρυξελών. Τα προσωπικά δεδομένα αποτέλεσαν αντικείμενο συλλογή ναι και ε, αντικείμενο αυτών των διαπραγματεύσεων. Επομένως, ε, τελικά, σε αυτή τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, προέβησαν κάποιοι ιδιωτικοί φορείς. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφιλείς πλευράς Βρυξελών και μελών και μόνος θα πρέπει να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να συμβουλήσουμε του Αμερικανού με μοναδικό να των ασφάλεια των πολιτών. Πρόεδρο. Κύριε Ζήστλα, μήπω δεχόσαστε ένα ερώτημα που θέλει να υποβάλει ε, ο κ. Αλφαρό. Κύριε Ζήλστρα, δεχόσαστε ερώτημα. Ναι, καλώς. Κύριε Άλβαρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσε να μου κάνει τη χάρη ο συνάδελφος να εξειδικεύσει τι εννοεί όταν λέει ότι ε, το Ισλάμ ε, είναι αιστεία ε, τρομοκρατικών επιθέσεων. έχετε το αυτό είναι παράδειγμα αφελίας. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι έχουμε χιλιάδες επιθέσεων από πλευράς Ισλαμιστών, τρομοκρατών, Λονδίνο, Δίδυμη Πύργη κλπ. Δεν λέω ότι το Ισλάμ η πηγή. Αλλά διαβάστε τι εφημερίδε. Η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι απαράδεκτη. Τι λέει, πρόκειται περί ψευδέστηση επόμενα. Είναι κάτι πολύ, πολύ στο για ασφάλεια των Καλώ για δύο λεπτά. Το επόμενο όνομα που έχω στον καταλογό μου είναι Βέμπερ, ο κ. Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκπρόσωπε του Συμβουλίου, θα πρέπει όλοι να δεχτούμε ότι όλους μας απασχολεί το θέμα της φύλαξης των δεδομένων. Ε, βεβαίως μας ενδιαφέρει η προστασία των πολιτών μας πάνω απ' όλα και επίσης ε, κοινό μας μέλημα είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα θύματα της Τουλούζης επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Κοινοβούλιο. Ε, όλα αυτά πρέπει να τα σταθμίσουμε. Η ομάδα ΕΛΚ θεωρεί ότι η ΕΠΑ στην μάχη κατά της τρομοκρατίας η ΕΠΑ λοιπόν στη μάχη αυτή είναι η συμμαχή μας, η εταίρη μας. Έτσι τους βλέπουμε και από κοινού θα θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους ε, αυτό το παιχνίδι ρόλων ότι οι Αμερικανοί είναι οι κακοί και συλλέγουν τα δεδομένα, οι Ευρωπαίοι όμως ωφελούνται από αυτή τη συλλογή, αυτό το παιχνίδι δεν θέλουμε να το παίξουμε. Από κοινού θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε και οι Ευρωπαίοι εμείς δράση. Ε, όλοι, ε, όλα τα κυρίαρχα κράτη έχουν το δικαίωμα να ζητούν προϋποθέσεις και στοιχεία για όσους εισέρχονται στο έδαφό τους και με την Αυστραλία έχουμε κάνει τέτοιε συζητήσει και με τον Καναδά και τώρα με τη ΣΥΠΑ. Η τωρινή συμφωνία συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Όσοι καταψηφίσουν την ε, συμφωνία θα έχουν λιγότερη ασφάλεια δικαίου. Αυτή είναι η τωρινή εναλλακτική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επίτροπο, διότι κατέστησε σαφές ότι από ε, ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρότερη και μπορεί να καταφέρει περισσότερα πράγματα από ότι 27 αν διαπραγματευτούν μεμονωμένα. Δεχόμαστε την εταιρική σχέση με τους Αμερικανούς, προσβλέπουμε στο μέλλον τη συζήτηση για συμφωνία πλαίσιο για την προστασία δεδομένων ε, τη λαμβάνουμε υπόψη και παρακαλώ τους Αμερικανούς στις διαπραγματεύσεις αυτές να ε, συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη τα ε, παγκόσμια, τα διεθνή ε, πρότυπα για την προστασία των δεδομένων. Αν εμείς ε, θεσπίσουμε δεδομένα από κοινού, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, στα πλαίσια μιας συμφωνίας πλαίσιο, αυτό θα αποβεί προς όφελος των πολιτών μας. Συνάδελφε Βέμπερ, υπάρχουν δύο συνάδελφοι που θα σε υποβάλουν ερωτήσεις. είστε διαθέσιμος να απαντήσετε. Ξεκινάμε με τον κ. Ταβάρεσου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βέμπερ, σε μια συζήτηση έχουμε κάθε υποχρέωση να είμαστε ρεαλιστές έναντι των πολιτών μας. Να μην δημιουργούμε πανικό. Κάνατε μια δήλωση, ε, είπατε αρκείτε να δείτε τι συνέβη στην Τουλούζη. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς συσχετίζεται αυτά που συνέβησαν στην Τουλούζη με τη συμφωνία. Γνωρίζαμε το ταξίδι στο Πακιστάν του τρομοκράτη της Τουλούζης τι θα έκανε ο συνάδελφος Βέμπερ, θα τον εμπόδιζε να ταξιδέψει ή αν υπάρχει τρόπος να εμποδίσει κανείς, μπορεί να εμποδίσει κανείς την Τουλούζη μέσω σώρευση αυτών στοιχείων, ο συνάδελφο έχει υποχρέωση να παραμένει στα όρια μια συζήτηση τεχνική και ραλιστικής και να μην χρησιμοποιεί φρικτά γεγονότα όπω αυτό τη Τουλούζη για να δημιουργεί πανικό στου πολίτε. Κυρίε συνάδελφε, ε, οποιοςδήποτε γνωρίζει ε, ζητήματα ε, ανακρίσεων θα απαντούσε ότι το ζήτημα είναι συνολικό. Δηλαδή πολλά πρέπει να ληφθούν υπόψη τηλεφωνικές επαφές τους, το, τις κινήσεις του υπόπτου. Υπάρχει μια συνολική εικόνα. Εγώ δεν είπα ότι ένα δεδομένο θα οδηγήσει στη σύλληψη. Είπα όμως ότι μας ενδιαφέρει η προστασία δεδομένων των πολιτών, αλλά πρέπει να σταθμίσουμε και αυτά τα οποία θα πρέπει να ε, ζητήσουμε ως δεδομένα, τι πρέπει να βρούμε, ούτω ώστε στο μέλλον να αποτρέπουμε τρομοκρατικά πλήγματα. Αυτό πρέπει να σταθμίσουμε. Πρέπει λοιπόν να ε, ε, σεβαστούμε το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν ορισμένα απαραίτητα δεδομένα. Συνάδελφε Άλμπρεχτ. Αξιότιμη κυρία Βέμπερ, σέβομαι την άποψή σας, αλλά ε, σκεφτόμενος αυτά που λέτε, ε, και όταν πρέπει να κάνουμε συμφωνίες και με τρίτες χώρες πώς αντιδράτε από, ε, στις, στα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας και της Κίνας που θα ζητήσουν παρόμοια πράγματα όταν παίρνουν τις σχετικές πληροφορίες οι Αμερικανοί. Γιατί να μην πάρουν και η Κίνα και η Σαουδική Αραβία ε, νόμιμα μέσα τις, τα στοιχεία αυτά μέσα από συμφωνίες με τη συμφωνή γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί και άλλα τέτοια μέτρα να μιμοποιηθούν από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, δέχεται οτιδήποτε αποφασίζουν τρίτες χώρες ανεξάρτητα από το αν αυτές συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή όχι. Ε, κυρία Άλμπρεχτ, όταν εγώ μιλώ με τις ε, διοκτικές αρχές, με ενημερώνουν ότι πολλές ε, προετοιμασίες τρομοκρατικών πληγμάτων στην Ευρώπη δεν θα είχαν προληφθεί αν δεν υπήρχε η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό λέω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εταίρος της Ευρώπης στην κοινή πάλι κατά της τρομοκρατίας. Αν θεωρώ ότι είναι δίκαιος εταίρος η είπα, τότε ευχαρίστω να καθίσω και να διαπραγματευτώ μαζί τους μια συμφωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εν λευκό επιταγή και, ε, όλες οι άλλες τρίτες χώρες. Ε, μπορεί να ε, ε, διαφοροποιούνται εδώ οι απόψεις μας. Εγώ θεωρώ ότι η ΕΠΑ είναι εταίρος και η Κομισιόν με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται και μπορεί να παρακολουθεί τους Αμερικανούς και να βλέπει πώς χειρίζονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα. Εγώ θέλω να είναι ισχυρή η Ευρώπη, αλλά δέχομαι ότι είναι και ένας τίμιος εταίρος η ΕΠΑ που θέλει μαζί μας να συνεργαστεί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Υπάρχει και τρίτη ερώτηση για σας. Σα ε, σας προτιμούν σήμερα. Ο κύριος Λάικφριτ έχει το επόμενο ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βέμπερ, σας γνωρίζω καιρό και σας γνωρίζω ως έναν αυστηρό υπέρμαχο του, κράτου δικαίου, του κράτους δικαίου. Εκπλήσωμαι λοιπόν ακούγοντας εσάς και την ομάδα σας ε, και τη θέση σας στη συζήτηση αυτή. Ε, λέτε ότι είστε υπέρ μια συμφωνία που για μένα είναι παράλογη. Λέτε ότι αν δεν υπήρχε η ΕΠΑ θα έκαναν ούτω ή άλλω ό,τι ήθελαν ανεξάρτητα από το τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό όμω είναι εκβιασμό, ε, κύριε Βέμπερ. Αν δεχτούμε, θα δεχτούμε δηλαδή τη συμφωνία επειδή φοβόμαστε ότι οι Αμερικανοί θα κάνουν ό,τι θέλουν έτσι κι αλλιώ. Μα δεν είναι δυνατόν. Πώ θα τα εξηγήσω όλα αυτά στου εκλογεί μου. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να πω στον κύριο Μορβάη ότι έχω δεχτεί τρεις ερωτήσεις γαλάζιας κάρτα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε και άλλες ερωτήσεις. Και διότι πρέπει να στη συζήτηση. Και μετά μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτησή σας και προ άλλον αγορητή. Η ερώτηση της παρανομίας μπορεί να κρυθεί πολιτικά. Εκεί οι απόψεις μας διαφοροποιούνται σε σχέση με τη συνθήκη. Ε, Υπάρχει όμως η Κομισιόν και η νομική της υπηρεσία που μας λέει ότι η συμφωνία είναι εντάξει. Αυτή είναι η νομική βάση. Αν άλλοι έχουν άλλη άποψη, αν συνάδελφοι διαφοροποιούνται, αν κράτη-μέλη διαφοροποιούνται, κυβερνήσεις στην Ευρώπη, τότε μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ε, σύστημα δικαίου. Το να ε, λέμε και να υπονοούμε ότι υπάρχει παρανομία ενώ η νομική υπηρεσία της Κομισιόν λέει ότι είναι εντάξει, ε, δεν είναι σωστό. Η, πώς θα ε, εξηγήσω με τα θέματα στους εκλογείς ε, πώς θα απαντήσετε εσείς στους εκλογείς σας όταν δεν υπάρχουν στα θέματα ανταλλαγής δεδομένων καθόλου κανόνες. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε συνάδελφο Λόπε Αγγιλάρ για δύο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, έχω την τιμή να προεδρεύω τη Επιτροπή των ε, Δημοκρατικών Ελευθεριών και ε, ει βάθο και επί πολύ εξετάσαμε το θέμα. Ήταν ε, αρκετά εντατική διαδικασία και επομένως με δημοκρατικές διαδικασίες η πλειοψηφία απεφάσισε όπως φαίνεται για το της ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ της συμφωνίας ούτως ώστε να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο τελικά για τη σύμφωνη συμφωνία και 23 ήταν κατά. Αυτό ήταν αποτέλεσμα επομένως των εργασιών της Επιτροπής μας κατά τις διαπραγματεύσεις γιατί θέλαμε πρώτα-πρώτα να περιχαρακωθεί αυτή η χρήση της συμφωνίας και έτσι και από την άλλη ε, πλευρά ε, να, ε, να περιχαρακώσουμε ποια εγκλήματα θα, θα καταπολεμηθούν και είπαμε ότι θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία επισύρουν ποινή πάνω από τρία χρόνια και έτσι ήμασταν πιστοί στις αρχές μας κόβεται το μικρόφωνο του ομιλητή και επίση κανονίσαμε το πόσο καιρό θα έχουμε την ε, ε, κατακράτηση των δεδομένων για κάποιο είδου εγκλήμων, εγκλήμων με τρομοκρατία για 15, την... θα γίνει αυτό 15 χρόνια. Και επίση είπαμε να έχουμε χρήση των δεδομένων με το σύστημα PUS ε, και να μην γίνεται δυσμενής διάκριση μέσω της χρήσης των στοιχείων. Επομένως έτσι και εμείς συμβάλαμε στην ε, αποκριστάλωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η εναλλακτική. Το να αφήσουμε το κάθε ένα από τα 27 κρατη να διαπραγματευτούν. Αυτό δεν θα κάνουμε τίποτα ισχυρότερη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήμασταν αντίθετα πιο ευάλωτοι. Αναγνωρίζουμε πάντως ότι από πρακτικής πλευράς οι πολίτες διέχονται τώρα από τη συμφωνία του 2007. Αυτό θα σημαίνει. Το οποίο δεν είναι καλύτερο. Θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Δεν θα είχαν περισσότερες εγγύσεις. Θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Επομένως, η λογική λέει ότι τώρα έχουμε μια βελτίωση. Έχουμε εγγύηση από πλευράς δικαίου, από πλευράς ισχυόντων νόμων. Και έτσι οι αεροπορικές εταιρείε. Οπότε, από τώρα και στο εξή και οι αεροπορικέ εταιρείε θα διέπονται από αυτό τη συμφωνία. Άλβαρο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε δεν ήταν εύκολη για τους φιλελευθέρους η απόφαση. Σταθμίσαμε πολλά επιχειρήματα, χωρίς δογματισμούς. Ίσως να είμαστε οι μοναδικοί σε αυτό το θέμα. Η ασφάλεια δικαίου, η σαφήνεια δικαίου, τα ξεκάθαρα λόγια είναι πολύ σημαντικά για τη συμφωνία. Ε, Υπάρχει κάποιο θέμα φύλαξης, το πεδίο εφαρμογής. Εδώ υπάρχει μια ανοιχτή ερμηνεία που δεν είναι πολύ σαφής. Ως ομάδα είμαστε υπέρ της ελευθερίας, της ελευθερίας του ατόμου. Ε, είναι πολύ σημαντικό εδώ να δούμε και την ανάληψη ευθύνης που έχουμε για την προστασία των πολιτών μας. Νομίζω ότι με την άρνησή μας ε, καθιστούμε σαφές ότι είμαστε κατά της υπονόμευσης της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ κύριε Άλβερο. Σαρτζεντίνη, επόμενο συνάδελφος. Κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν στην Τουλούζη οι προηγούμενοι αγορητές και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στους Νιγηριανούς που ήρθαν στο Άμστερνταμ για έναν Νιγηριανό που ήρθε στο Άμστερνταμ και μετά πήγε στο Ντιστρόιτ. Και υπήρχαν ε, πληροφορίες ότι έκανε κάτι παράνομο και είχαν και οι Γάλλοι πληροφορίες. Έχουν οι δυνάμεις ασφαλείας πληροφορίες για τα διάφορα άτομα και πρέπει να μπορούν να τα χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία. Καμιά φορά δεν χρησιμοποιούν σωστά τις πληροφορίες. Αυτό πρέπει να πετύχουμε για να αυξήσουμε την ασφάλεια. Δηλαδή, οι υπηρεσίες μας ασφαλείας να κάνουν ό,τι μπορούν με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Το PNR είναι ένα σύστημα που στέλνει ένα μήνυμα. Δείχνει την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Καμιά φορά τα παίρνουμε μια λογική απόφαση δεν υπάρχει τρόπος να επαναχωρήσουμε. Λοιπόν, αν συλλέγονται όλα τα στοιχεία αυτά για κάποιον που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, δεν είναι το σωστό μήνυμα που αποστέλουμε, ούτε είναι αποτελεσματικό τρόπο για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Σα ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ καταπληκτική αυτή η συζήτηση και όμω ε, εκεί που χάθηκε ε, το, το, το, το, το, νήμα ε, τη εκλογική είναι το τι έγινε πριν από 10 χρόνια που είχαμε πάνω από 10.000 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους της ΕΙΠΑ και κάποιος ο οποίος ε, τότε ε, ασχολείται με τις μεταφορές έλεγε ότι θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα ασφάλιση, ασφάλειας για να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη και ακριβώς είπαμε ότι είναι ε, πάρα πολύ απέσια αυτή η επίθεση, να την αντιμετωπίσουμε και επομένω και εγώ θεωρώ ότι θα ήταν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εάν η κυβέρνησή μου δεν θα έκανε ό,τι πρέπει για να με εξασφαλίσει την, την, την, ασφάλειά μου όταν ταξιδεύω στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκτός της χώρας. Ε, πολλές φορές θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα τα οποία είναι σκληρά, αλλά τελικά είναι θέμα στάθμισης των πάντων. Και επομένω θα πρέπει να πούμε στην εισηγήτρια ότι στα 37.000 πόδια δεν τους καίγεται ε, καρφί των τρομοκρατών για τα, για, ε, για τα ερωτήματα για τις αμφιβολίες αυτές, τον προβληματισμό. Εγώ έχω δουλεύει τόσα πολλά χρόνια σε αεροπορική εταιρεία και, και, και, και, ξέρω τι γίνεται στους τρομοκράτες. Από τη δεκαετία του 70 δεν γνωρίζουν όρια, δεν γνωρίζουν ηθικούς ε, φραγμούς και συνήθως ούτε καν χρειάζονται αιτιολογία για να αφαιρέσουν ανθρώπινε ζωέ. Απλώ θέλουν να κάνουν για δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη εντύπωση, θέλουν ένα μήνυμα. PNR. Τι πάνω από PNR. Είναι κάποιε πάρα πολύ βασικέ στοιχειώσει Ε, δεν είναι και, και τίποτα τρομερό. Οπότε γι' αυτό σα λέω, Πρόεδρε, και εγώ και οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, κάνουμε σκληρέ διαπραγματεύσει, τόσο ώστε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των ε, πολιτών τη Ένωση και όλων. Ε, ούτω ώστε να υπάρχουν ε, κάποιε εγγύσει. Είναι πάρα πολύ σημαντική επομένω αυτή η πληροφορία και επομένω η ήδη για ε, τι απόπειρε στο Λονδίνο μπορέσαμε επομένω να, έτσι να διώξουμε εγκληματίε παντού. Οπότε παρακαλώ συνάδελφοι να επιψηφίσετε αυτή τη συμφωνία. Ε, έγινε διαπραγματεύσει, καταλήξαμε σε μια λογική συμφωνία και έτσι οι Βρετανοί και όλοι οι Ευρωπαίοι πρόκειται να ε, έχουν ασφάλεια όταν ταξιδεύουν. Κυρία Φώστα, σα ευχαριστώ. Δεχόσαστε ερώτηση από πλευράς της κυρίας Ιντεβέλτ. Yes. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφο Φώστερ το εξή. Περιφρονεί και εμένα και τους άλλους αντίθετη συμφωνία λέγοντας ότι δεν έδωσε επαρκή σκέψη στην ασφάλεια. Ήθελα να ξέρω, διαβάσατε τη συμφωνία και τις αντιρρήσεις κατά αυτής και απαντήσατε στην ερώτηση. Πώς η δημόσια υγεία, η μετανάστευση, και το ελληνικό έλεγχο, οι σχετικέ πολιτικέ επηρεάζουν την πορεία των αεροσκαφών στα 37.000 πόδια, όταν ύπτανται στα 37.000 πόδια. Απάντηση. Δεν νομίζω ότι περιφρονώ την εισηγήτρια ή, α, ή την υποτιμώ. Ε, νομίζω ότι τώρα θεωρεί ότι γνωρίζει τα πάντα η την υποτιμω νομιζω οτι τωρα θεωρει οτι γνωριζει τα παντα η τρομοκρατια και αυτό πιστεύω. Ήμουν συνάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε οργανώσει ο κύριος Κέρχοπ με αξιωματούχους του Υπουργείου ε, Εσωτερικών και δόθηκαν πληροφορίε η κατάσταση βοηθούσε την έκθεση. Μετά από 10 χρόνια, κυρία εισηγήτρια, κάποια από τα σχόλια που μα ε, εκφράσατε σήμερα το πρωί θεωρώ ότι είναι εντελώ αφέλη. Νομίζω ότι ζείτε καμία φορά σε άλλο πλανήτη. Θεωρείτε ότι έχετε το μονοπόλιο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια δεν έχετε το μονοπόλιο. Οι υπόλοιποι εδώ σε αυτή την αίθουσα πιστεύετε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματά μα και να διατηρούνται με ασφάλεια τα στοιχεία μα. Βεβαίω δεν είμαστε ανόητοι, δεν χρειαζόμαστε μαθήματα από ανθρώπου σαν και εσά. Αλλά αυτό που εξίσουμε γνωρίζουμε είναι ότι οι κυβερνήσει μα και οι πολιτικοί μα θα πρέπει να λάβουν σκληρέ αποφάσει καμιά φορά και δεν είναι πάντα εύκολο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη συμφωνία που έχουμε μπροστά μα. Πολύ σοβαρέ ήταν οι διαπραγματεύσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα συνεχίσει πολύ καλά την πορεία τη που έπρεπε. Κυρία Φόλστερ, μην βγάζετε τα ακουστικά σα, βάλτε τα ακουστικά σα παρακαλώ. Υπάρχουν άλλε δύο ερωτήσει ε, που θέλουν να υποβάλουν. Από πλευρά και από πλευρά Άλμπρεχτ. Να πω στους συναδέλφους ότι αυτό το εργαλείο της γαλάζιας κάρτας είναι πολύ χρήσιμο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με, κάποια, ε, με κάποιο έλεγχο. Διαφορετικά ο χρόνος των συζητήσεων ε, θα εξαντληθεί. Μορμπάι. Μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτηση σας κύριε Μορμπάι. Ε, Ευχαριστώ. Με κάθε σεβασμό να ρωτήσω κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, περιμένετε να τελειώσω, θα συμφωνούσατε ότι μια κυβέρνηση η δική μας ή κάποια άλλη δεν έχει καμιά δουλειά να ανακατεύεται στο πότε ταξιδεύουμε, με ποιους, πόσο συχνά, ε, πόσα χρήματα δίνουμε για το εισιτήριο ε, ή αν ε, έχουμε ε, κάποια προβλήματα υγείας κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Βέβαια η κυβέρνηση μπορεί να έχει νόμιμο συμφέρον να συλλέγει δεδομένα αν πρόκειται να προστατεύσει ζωές μέσα από τις πληροφορίες αυτές και χάρη σε αυτές. Αλλά πώς ακριβώς θα προστατευθούμε από την τρομοκρατία μέσα από αυτή την προστασία των δεδομένων μέσα από αυτή τη συλλογή δεδομένων και την ε, μείωση της προσωπικής μας σφαίρας. Συνάδελφοι, παρακαλώ να περιοριστείτε στο διαθέσιμο χρονικό διάστημα. Εντάξει, δέχομαι το σχόλιά σας. Οι αεροπορικέ εταιρείε πάντοτε συνέλεγαν δεδομένα δικά μα εδώ και δεκαετίες όταν κάναμε κράτηση εισιτηρίων. Ε, είναι πολύ λίγο διαφορετικές οι πληροφορίες από αυτές που συλλέγονταν πριν από την 11η, 9η Σεπτεμβρίου. 11η Σεπτεμβρίου. Ε, Πόσες είναι υπερβολικά πολλές πληροφορίες. Το πρόβλημα είναι ότι οι, τρομοκρατίες, οι τρομοκράτες δεν σταματούν στα σύνορα. Η τρομοκρατία είναι διεθνής. Πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε πληροφορίες που δεν θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε. Και είναι δύσκολο οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί να ε, πουν... Ε, ότι είναι προς το συμφέρον μας να το κάνουμε αυτό. Ε, δεν υπάρχει μια άμεση απάντηση. Είναι σορευτική, με βάση σορευτικά στοιχεία η απάντηση που δίνεται και με βάση την, προ, ε, την πρακτική των τρομοκρατών. Ε, ο κύριος Άλμπρεχτ, κυρία Φώστερ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ε, λέτε ότι τα στοιχεία PNR είναι βασικές πληροφορίες, λίγες πληροφορίες. Γνωρίζετε ότι με την ε, πληροφόρηση API το κομμάτι της βασικής ε, πληροφόρησης διαβιβάζεται διεθνώς αυτομάτως όταν δηλαδή μιλάμε για στοιχεία σχετικά με το ποιο ποιος βρίσκεται σε ποιο αεροπλάνο. Επίσης ε, αναφέρεται το τι θα αγοράσω με την κάρτα επιβίβασης ε, στα καταστήματα φορολόγητων, ε, παρακολουθείτε η πιστοτική μου κάρτα. Ε, όλα αυτά ε, συμπεριλαμβάνονται και στις έρευνες και στις περαιτέρω αναλύσεις λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη. Κοιτάξτε κύριε Άλβεχ, μιλήσατε 15 φορές σήμερα το πρωί. Σεβαστούμε και του άλλου συναδέλφου που είναι παρόντες και είναι εγγεγραμμένοι να πάρουν το λόγο. Κυρία Φώστερ, απαντήστε, ε, αλλά παρακαλώ τηρήστε το χρονικό διάστημα που σας είναι διαθέσιμο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, η απάντηση είναι ναι. Πολύ καλά. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ο κ. Μποργέζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν να προχωρήσουμε στο θέμα, υπάρχει, πρέπει να υπάρχει συζήτηση ισορροπία Υπόθηκαν σωστά πράγματα λοιπόν και θεωρώ ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση. Και δεν υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις βάσιμες. Σήμερα το πρωί, αντί να μπούμε στη φιλοσοφική συζήτηση, όσον αφορά το δίκαιο, θα πρέπει υπεύθυνα να εξετάσουμε το δίκαιο στην ασφάλεια για τους συμπολίτε μας. Κυρίως για εκείνους τους νέους, τους εργαζόμενους που ήταν θύμα της τρομοκρατίας, που έπληξε και ένα τρένο που μετέφερε τους εργάτες, τους νέους, το χάρη, και ούτω καθεξής. Και το δικαίωμα στην ασφάλεια, που πρέπει να επικρατεί ακόμα και σε προσωπικές και πολιτικές θέσεις. Μια ομάδα ευρωσκεπτιστικής που δεν πιστεύω ότι μπορεί, όπως είπε ο κ. Μπάτε, να ψηφίσει. Και όσον αφορά τη Λέγκα του Βορρά, σίγουρα θα υπερψηφίσει. Όχι διότι δεν θεωρούμε ότι είναι σημαντική η privacy, αλλά επικρέμεται διάχυτος ο τρόμος, η απειλή της τρομοκρατίας που μπορεί να είναι και πυρηνικής φύσεως. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μάλτσαρ. Η συμφωνία PNR αναμφίβολα δεν προστατεύει επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων διότι διαβιβάζονται τα στοιχεία και στη ΣΥΠΑ και στις τρίτες χώρες. Επίσης θεωρείται εκτελεστική συμφωνία στη ΣΥΠΑ. Το Κογκρέσο δεν την επικυρώνει, οπότε δεν είναι και νομικά δεσμευτική συμφωνία για τη ΣΥΠΑ. Όταν ε, παρουσιάζονται στοιχεία για τις ε, ε, ταξιδιωτικές κινήσεις όλων των πολιτών Πώς θα μπορούσαμε, είναι απλοϊκό να θεωρήσουμε ότι χωρίς δεσμευτική συμφωνία μπορούμε να παρέμβουμε στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων. Ε, αναφέρθηκε, ε, νομίζω ότι θα έπρεπε η Κομισιόν να επεξεργαστεί μια καλύτερη συμφωνία για του πολίτε τη. Ευχαριστώ κύριε Μόντσορ. Κύριε τέλεια δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ο πυρήνα του θέματο, όταν ψηφίσουμε, θα είναι εξή. Θα πρέπει να απαντήσουμε στην ερώτηση. Αυτή η συμφωνία πετυχαίνει σωστή ισορροπία μεταξύ εξίσου σημαντικών στόχων που όλοι μα ε, θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, προστασία των πολιτών μα, ασφάλεια δηλαδή από την μια πλευρά και προστασία τη ιδιωτική ζωή από την άλλη. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κρίνουμε ε, τη συμφωνία που έχουμε μπροστά μας πριν μπορέσουμε να πούμε ναι ή ου. Η απάντησή μου σε αυτό το ερώτημα είναι ναι. Νομίζω ότι πετυχαίνουμε μια σωστή ισορροπία με αυτή τη συμφωνία παρόλο που είμαι ο πρώτος που δέχεται ότι αυτή η συμφωνία δεν αντιστοιχεί πλήρω στι υψηλές μας προσδοκίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και δεν αποτελεί το, τη σημαντική πρόοδο που θέλουμε να πετύχουμε. Έχω τρει λόγου για του οποίου πιστεύω ότι θα έπρεπε να υποστηρίξουμε τη συμφωνία. Οι περισσότεροι λόγοι ήδη αναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα, έχοντα αυτή τη συμφωνία είναι κάτι καλύτερο από το να μην την έχουμε καθόλου. Και για λόγου ασφαλεία, αλλά και για την ιδιωτική ζωή των πολιτών για την προστασία τη. Αυτή η συμφωνία παρέχει καλύτερο πλαίσιο προστασία των δεδομένων από ότι η παρούσα συμφωνία του 2007 και ενδεχομένω και οι διμερεί συμφωνίε οι οποίες θα έπρεπε να ισχύουν άνευ της παρούσης. Και άνευ αυτή της συμφωνίας τα στοιχεία όπως αναφέρθηκε θα εξακολουθούν να αραίουν χωρίς μέτρα διαφύλαξης. Δεύτερον, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία από τα άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν και μεταβούν εκεί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι δυνατόν να προστατεύσουν τη ιδιωτική του ζωή όταν επιλέγουν να το κάνουν αυτό. Στην πράξη, Χωρίς αυτή τη συμφωνία ίσως ε, καταλήξουμε με παρεμπόδιση της εναέριας, των εναέριων ταξιδίων μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τους επιβάτες και πιο χαμηλή προστασία των ιδιωτικών στοιχείων. Σίγουρα η επεξεργασία στοιχείων PNR βοηθά πράγματι την ασφάλεια των πολιτών μας δεν θα πρέπει να αποτελεί ταμπού στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι η προστασία των πολιτών μας είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Ναι, πόρα απέχει από το να είναι τέλεια συμφωνία, αλλά τελικά όμως είναι καλύτερη η θέση των πολιτών μας με αυτή τη συμφωνία παρά όχι. Κύριε Μπουσετήλ, δεχόσαστε πλευράς ο Ρομέρο ένα ερώτημα. Ορίστε. Κύριε Μπουσουτήλ. Γνωρίζετε ότι στα εθνικά κοινοβούλια έχουμε στο επίπεδο Μόνο τρεις χώρες έχουν ε, κατοχυρώσει το PNR στην εθνική νομοθεσία. Και, το χρησιμοποιούν κατά τη μετανάστευση ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία και η Δανία που είναι η τρίτη χώρα και το έκαναν. Μόνο, μόνο, μόνο το, το, το χρησιμοποιούν για περιπτώσεις τρομοκρατίας. Γνωρίζετε ότι τώρα προσκρούμε στι αρχές τόσων εθνικών κοινοβουλίων και πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως γνωρίζετε και έχουμε επίσης ε, ε, το κείμενο της Κομισιόν δεν είναι το μόνο το οποίο έχει συνταχθεί πάνω σε αυτό και δεν είναι μόνο νομικοί αυτοί που τα συνέταξαν αυτά τα κείμενα έχουμε επίσης και κάποιους επόπτες των ε, κρατών μελών οι οποίοι ε, οι έχουν ε, συντάξει εκθέτη τη μία εκθέτω την άλλη και βεβαιώνουν εκεί ότι αυτή η συμφωνία προσκρούει στι αρχέ κατοχή των δημιουργικών δικαιωμάτων. Μπορούσε ότι ναι, το γνωρίζω αυτό, Πρόεδρε. Επίση γνωρίζω ότι ε, θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η συμφωνία για τη κατοχή τη τρομοκρατία και γι' αυτό και θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το βασικό ε, ψεγάδι σε αυτού οι οποίοι συμφωνία ε, λένε ότι δεν προστατεύεται ο δυτικό βίο. Το θέμα όμω, το πρόβλημά του είναι ότι δεν βλέπουν ότι χωρί τη συμφωνία τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Θα είχαμε ακόμα λιγότερε εγγύσει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οπότε παρακαλώ, όσοι δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία, α λάβουν υπόψη αυτό το σημαντικό στοιχείο που προανέφερα τώρα. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφε Σίπελ, έχετε το λόγο για δύο μισή λεπτά, κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τρομοκρατικά πλήγματα πριν από χρόνια έδωσαν ένα, έναυσμα για τη φύλαξη δεδομένων. Η τρομοκρατία όμως δεν αρκεί για να νομιμοποιήσει τη φύλαξη δεδομένων ε, απέναντι στους πολίτες. Γι' αυτό μιλάμε για οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα, εμπορία ανθρώπων Εκατομμύρια στοιχεία ε, συλλέγονται με περιορισμένες επιτυχίες. Η κυρία Μάλμσον λέει ότι η προστασία δεδομένων βελτιώθηκε και λέει ότι κάποια δεδομένα ε, τώρα μόνο 10 χρόνια φυλάσσονται. Όμως η προστασία δεδομένων αρχίζει νωρίτερα με το συγκεκριμένη στοχοθέτηση ή τον περιορισμό των σχετικών δεδομένων. Τι γίνεται όμως με το, την παρούσα συμφωνία και το κείμενο της εκατομμύρια δεδομένα ε, αθώων πολιτών φυλάσσονται για τουλάχιστον 10 χρόνια, επί 10 χρόνια ε, επανεξετάζονται και την χάνουν επεξεργασία για διάφορους σκοπούς. Ε, αφορούν αδικήματα με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια πρέπει να ληφθεί υπόψη για αδικήματα για τα οποία εδώ ε, δεν γίνεται καν δίκη στις ΗΠΑ η ποινή είναι πολυετής φυλάκιση. Τα αδικήματα πρέπει να είναι διασυνοριακά. Ε, βεβαίως... Ε, ε, αυτό ισχύει για όλους εμάς που βγάζουμε εισιτήρια με επιστροφή. Ε, υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων προς άλλες αρχές και προς άλλα κράτη. Αυτό δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις και είναι κρίμα που η αξιολόγηση μέχρι τώρα δεν προβλέπει προστασία δεδομένων ε, απέναντι σε αυτές τις χώρες. Επίσης ε, υπάρχουν ε, στις ΗΠΑ άνθρωποι που κατηγορούνται για τρομοκρατία και παραμένουν προφυλακισμένοι για πολλά χρόνια μεταξύ αυτών και αθώοι. Θα πρέπει η τρομοκρατία να καταπολεμηθεί αλλά εδώ πάμε πολύ μακριά. Όλους τους θεωρούμε υπόπτους τους ε, ε, παραδίδουμε στις ΗΠΑ αντί να προστατεύσουμε εμείς τους πολίτες μας και τα δικαιώματά τους. Ο κύριος Άλμπρεχτ ρώτησε αν ε, πρέπει να ντρέπονται αυτοί που ψηφίζουν υπέρ. Όχι, κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται για την τωρινή του απόφαση, αλλά ανησυχώ βαθύτατα για την κατεύθυνση που ακολουθούμε εγκρίνοντας τη συμφωνία. Και γι' αυτό είμαι βαθύτατα πεπισμένη ότι πρέπει να καταψηφίσω. Συνάδελφε Γκρίσμπεκ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το SWIFT, το ACTA, το PNR είναι ακρόνημα που συνήθως πολύ συχνά αναφέρονται και ανησυχούν τους Ευρωπαίους που δεν γνωρίζουν πραγματικά τι κρύβεται πίσω από αυτά. Ε, ποια πραγματικότητα κρύβεται. Εποπτεία, πολύ γενικευμένη όσον αφορά τους επιβάτες, μια συμφωνία από οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν πάρω το αεροπλάνο, θα γνωρίζουν τι θέλω να φάω, ποια είναι η συμπεριφορά μου στο αεροδρόμιο, στοιχεία όσον αφορά την υγεία μου κλπ. Χωρί να αναφερθώ σε όλα τα επιχειρήματα που ήδη αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί σε μια συζήτηση ζεστή, μα θερμή. Θα ήθελα να Θέλαμε να ζητήσουμε από, την δεκαετία, από το 2007 εγγυήσει όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές που θα θέταμε, που θα μας επέτρεπαν να πετύχουμε μια συμφωνία του Κοινοβουλίου. Σήμερα δεν έχουμε αυτούς τους όρους όσον αφορά την αμοιβαιότητα, ούτε όσον αφορά την αναλογικότητα, όπως το υπενθύμησε ο έξοχος συνάδελφος Γκρέαμ Βάτσον όσον αφορά τη θέση των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Ή αυτά που είπε η κυρία Φόρστε τα οποία αφισβητώ, λέγοντας ότι δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά στο PNR. Αν δεν, ζητάμε πολλά, αν δεν υπάρχουν πολλά στο PNR, θα ζητήσουμε αμοιβαιότητα από τη ΣΥΠΑ. Αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να πάρουμε, ότι θα πάρουμε τίποτα περισσότερο, θα πετύχουμε περισσότερο. Πρέπει να ζητήσουμε από τους ε, δικαστέ να κρίνουν. Δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε τι ευθύνε μα. Πρέπει να δημιουργήσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θέλουμε ασφάλεια, κατά πολέμηση τη τρομοκρατία και από την άλλη πλευρά διαφύλαξη των ελευθεριών. Και γι' αυτό θα καταψηφίσω αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Κυρία Φότχ, έχει το λόγο. Ναι, μετά από την αρχή της συζήτησης δεν υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία κατά κάποιο τρόπο δεν πλήττει τα δεμελιώδη δικαιώματα. Μερικοί απλώ λένε ότι είναι κάτι καλύτερο από το τίποτα, θα ήταν χειρότερα χωρί συμφωνία και τελικά ε, το να τρώνε λίγο τα δικαιώματά μα, αν πετυχαίνουμε κάτι όσον αφορά την ασφάλεια, μπορούμε κάτι, να, κάπου να καταλήξουμε. Αυτά αναφέρθηκαν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μια πολιτική καταπολέμηση τη νομοκρατίας για να είναι αποτελεσματική, όχι για να είναι μόνο ηθική, ή ότι για να συμμορφωθούμε για τι διεθνεί υποχρεώσει. Για να αποτελεσματική ε, πρέπει να σέβεται τα διεθνέ δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι υποχρεώσει μα. Και είναι ένα δικαστήριο μπορεί να διαλύσει ίσω αυτή τη συμφωνία. Πρέπει να απομισθούμε τι πολιτικέ μα ευθύνε. Γνωρίζουμε γιατί όπω είμαστε στο παρελθόν, οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν μπορούν να βασιστούν παρά μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα. Θα είμαστε στο πλευρό των πολιτών ή θα αφήσουμε να εντυπωσιαστούμε από απειλέ. Διότι το παρελθόν μιλά στην περίπτωση του συστήματο που δημιούργησε η CIA με τι μυστικέ φυλακέ, παράνομε μεταφορέ, βασανιστήρια στην επικράτειά μα. Ποιον θα βρούμε στο πλευρό μα στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξαγωγή των ερευνών και την εξέβρεση των υπευθύνων. Κανέναν. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Δεν έχουμε κανέναν μηχανισμό ελέγχου όταν οι υπηρεσίε βγαίνουν από το νομικό πλαίσιο και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Συνάδελφε Ρένα Άουζερ, θέλετε να δεχτείτε ε, μια ερώτηση από πλευράς της κυρίας Φώστερ. Κυρία Φλότχα. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για να σα πω κάτι για αυτό που η κυρία Φλότ μα είπε ότι όλοι οι πολίτε είναι κατά. Οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα αυτό το οποίο θέλουν ε, οι πολίτε είναι να εξασφαλίσουν την ανάληψη ευθύνη από τι κυβερνήσει του, όταν μετακινούνται και θέλουν να μετακινούνται ελεύθερα εντός και εκτός συνόρων. Θέλουν επομένω κάποιο να λάβει την ευθύνη για την ασφαλεία τους. Πρόκειται περί δυσκόλων αποφάσεων και οπότε ε, Ξέρετε τι, τι, τι, τι, τι, τι οι πολίτε και είδατε τι γίνεται με τι γαλλικέ εκλογέ. Δεν έχουν ιδέα, δεν ενδιαφέρονται για το PNR. Απλώ προσδοκούν από του πολιτικού να του ασφαλίσουν την ασφαλή μετακίνηση. Αυτό, το περιμένουν. Παρακαλώ, θέλετε να απαντήσετε. Κανένα δεν αρνείται όμως ότι τώρα υπονομεύονται τα δικαιώματα και λέτε ότι δεν ξέρουν. Αλλά τα, ε, αυτό το κάνει πράγματα ακόμα χειρότερα. Οπότε, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα χειρότερη παραγωγή των δικαιωμάτων το να μην ξέρουν τι έλεγχο γίνεται. Οπότε ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ε, αυτή, αυτή τον τρόπο ε, αντιμετώπισης τρομοκρατίας αλλά αμερικανικά οπότε έχουμε τις φυλακές, τα δικαστήρια, την αμερικανική μέθοδο, επομένω κάνετε λάθο κύριε Φώστα. Συνάδελφε ähm, Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 εψήφισε δύο ψηφίσματα κατά πλειοψηφία και διατύπωσε σαφείς όρους Τώρα η συμφωνία αντιβαίνει προς αυτές. Πρώτον, το profiling εξακολουθεί να μην αποκλείεται. Ήδη η μέθοδος pool εξακολουθεί να είναι δυνατή. Τρίτον, ο στόχος ε, περαιτέρω διαβίβασης δεδομένων δεν ε, ε εξειδικεύεται. Επίσης ο σκοπός ε, για τη μαζική φύλαξη δεδομένων δεν αιτιολογείται και η Κομισιόν δεν φρόντισε για εναλλακτικέ. Γενικά Καταλήγομαι ότι σε σχέση με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν σοβαρές δηλαδή ε, αντιφάσεις μεταξύ της συμφωνίας και αυτών των κειμένων και δικαστικών αποφάσεων. Ευχαριστώ συνάδελφε Μάουρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Η πτυχή, η εύθραυστη που όλοι οι συνάδελφοι και εκείνοι που θα υπερψηφίσουν ακόμα σήμερα κατήγγυλαν όσον αφορά τη συμφωνία είναι εύκολα, κάτι εύκολα κατανοητό αν αναφερθούμε σε κάτι που ανέφερε η κυρία Μάλσουμ και το Συμβούλιο. Αναφέρθηκαν με σαφήνεια σε νέε σημαντικέ παραχωρήσει ε, που, παρα, που στη συμφωνία. Παραχωρήσει. Η στάση αυτή της παραχώρηση είναι διαφορετική από την τοποθέτηση της αναγνώρισης των προνομίων των δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Είναι περισσότερο πολιτισμικό από ότι πολιτικό που αφορά τη σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των αμερικανικών αρχών. Και αυτό το πρόβλημα επέτρεψε αμερικανικές αρχές αντί να, να μόνο με τις διαπραγματεύσεις με τα κάτι μέλη να, να έρθουν σε επαφή με κάθε κάτος μέλος ε, ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζοντας την αντικειμενικότητα αυτού του γεγονότος, πιστεύω ότι όχι μόνο ανησυχία για την ασφάλεια, αλλά και το θέμα των προόδων που έχουν επιτευχθεί στην συμφωνία θα έπρεπε να μας οδηγήσει στην υπερψήφιση. Διότι ειλικρινά και η ενωμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οικοδομείται μία ανοιχτή. Δεν καταρφώνουμε με ένα μόνο κείμενο να μεταφέρουμε τη δυνατότητα να να... Ε, του να εμπιστευόμαστε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε καθημερινά. Πολύ σωστά το ανέφερε κύριε Αγγιλάρ ε... περιγράφοντας πόσο ζωηρή και βαθιά ήταν η συζήτηση στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Γι' αυτό η Ιταλική Αντιπροσωπεία του, του ΕΛΚ θα υπερψηφίσει ε, αυτή τη συμφωνία τους καλύτερους καιρούς. Ευχαριστώ κύριε Μάουρο. Γκόνς, συνάδελφος Γκόνς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και με το SWIFT, έχει δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχτεί τη συμφωνία. Όμως, το πρώτο είναι ότι δεν είχαμε αρκετή ενημέρωση. Ούτε λήθησαν υπόψη οι προϋποθέσεις που έθεσε το Κοινοβούλιο και οι όροι που έθεσε κατά τις διαπραγματεύσεις. Έγινε συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά έλαβε υπόψη κάποιες από τις προτάσεις μας. Πάντως συνεχίζω να πιστεύω ότι παρά το ότι επιδέχεται βελτιώσει αυτή η συμφωνία θα πρέπει να πούμε ναι σε αυτήν. Εάν δεν έχουμε αυτή τη συμφωνία τότε δεν θα έχουμε μια ενιαία ρύθμιση. Ούτε θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ε, πορεία και την τύχη των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, τα κράτη-μέλη σε διμερείς συμφωνία θα είναι αδύναμα έναντι τον ΗΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορεί το Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενημερώνεται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Και θα πρέπει αν χρειαστεί να ξαναδιαπραγματευτούμε. Επίσης, θα πρέπει οι επιβάτες να ξέρουν τι το προς δεδομένα. Έτσι θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Το ίδιο θα ισχύει βέβαια και έναντι των αεροπορικών εταιριών της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθήσει το πώ θα εφαρμοστεί η συμφωνία, το πώ χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και θα πρέπει να αναφέρει σχετικά στο Κοινοβούλιο, αν διαπιστώσει ότι δεν προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων. Και να ξαναρχίσει τη διαπραγματεύση că uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να δέχεται διαφορετικές απόψεις και πιστεύω ότι όλοι αντιμετωπίζουμε το κίνδυνο της διεθνούς τρομοκρατίας και διάφορους κινδύνους παγκοσμίου. Είναι κίνδυνοι παγκόσμιοι, χρειάζονται μια παγκόσμια απάντηση. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο και γι' αυτό καταλήξαμε σε διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη συμφωνία. Μπορεί να μην είναι τέλεια, όπως υπόθηκε, όμως ε, προσφέρει μια βεβαιότητα, εχέγγυα, για το σεβασμό διαφόρων δικαιωμάτων. Συμφωνώ ότι τα στοιχεία τα προσωπικά θα πρέπει να προστατευτούν. Οι πολίτες όμως έχουν και το δικαίωμα της ασφάλειας των προσωπικών του στοιχείων. Θεμελιώδης δικαίωμα εμπεριέχονται εγγυήσεις στη συμφωνία. Το ότι μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να εποπτεύουμε είναι καλό. Και εμπιστεύομαι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αμερικανικές Αρχές. Όλα αυτά είναι επιχειρήματα υπέρ της συμφωνίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η συμφωνία μας δίνει ένα, με το ένα χέρι κάτι και αποσύρει με το άλλο. Λέμε ότι τα στοιχεία δεν θα αποθηκεύονται πάνω από ένα εξάμεινο αλλά μπορούν ε, να ανακτηθούν και επί 15 ετία περισσότερο χρονικό διάστημα. Μπορούν να γίνουν δικαστικές προσφυγές, αλλά οι Αμερικανικές αρχές δεν μας επιτρέπουν προσφυγή σε δικαστήριο αν υπάρξει κάποια παράβαση. Και αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε κάποιες περιστάσεις. Αυτή η συμφωνία ίσως ακυρωθεί σε κάποιο δικαστήριο. Αν όμως Θέλουμε μια συμφωνία για την οποία δεν υπάρχουν εγγυήσεις έναντι δικαστικών προσφυγών, δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Για την ώρα υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη. Έλλειψη αξιοπιστίας έναντι των πολιτικών. Μας λένε ότι δεν προστατεύουν τους πολίτες. Η κυρία Φώστερ μας λένε ότι δεν ξέρουν οι πολίτες τι σημαίνει το PNR. Και μπορούμε, μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο οι πολίτες. Όμως αν το δεχτούμε αυτό θα χάσουν κάθε, ε, πολιτικ, κάθε αξιοπιστία όσον αφορά πολιτικούς. Κύριος Μπόστ, έχετε ένα ερώτημα να υποβάλει. Μία ερώτηση. Πώς βλέπεις την εναλλακτική, δηλαδή αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία θα γίνεται συλλογή δεδομένων στη ΣΥΠΑ, ανεξέλεγκτα όμως και κατά πάσα πιθανότητα ε, η, η ελευθερία των πολιτών θα είναι στέκονται στις ουρές. Γιατί γιατί δεν θα επιδηλωθεί η κατάσταση των πολιτών που θα θέλουν να ταξιδέψουν στη ΣΥΠΑ. Δεν θα πρέπει να φροντίσουμε για τη βελτίωση της κατάστασης ε, των πολιτών να ταξιδεύουν και όχι να, τη χειροτέρεψη. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσο θα νομιμοποιήσουμε κάτι που παραβιάζει τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ομοθεσία την προστασία των δεδομένων. Όμως οι Αμερικανοί ήδη έχουν αυτά τα στοιχεία στην επικράτειά τους. Δεν μπορούμε όμως να νομιμοποιήσουμε αυτό που γίνεται. Γιατί αν το κάνουμε αυτό θα τεθεί ένα ερώτημα σε μερικά χρόνια. Θα κάνουμε και το ίδιο με την ε, Σαουδική Αραβία, τη Λατινική Αμερική, τη Ρωσία ή άλλες χώρες που και αυτές προσπαθούν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Κυρία Φώστερ έχει ένα ερώτημα, το δεχόσαστε. Ναι, λέει αγορητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω στον τελευταίο μιλητή ότι αν θέλετε να παραθέσετε αυτά που, είπατε, που είπα να είστε ακριβείς. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είπα αυτό που είπατε όσον αφορά την κατανόηση των πολιτών στο αφορά το PNR. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φτηνά ε, μέσα, ας βγούμε έξω. Αν αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε σαν πολιτικό επιχείρημα, δεν έπρεπε να καθόσαστε εκεί που καθόσαστε, αν αυτό είναι το καλύτερο σας όπλο. Επόμενο αγορητή. Κυρία Φώστερ, με τα χαρά σα απαντήσω. Σωστά σας παραθέσω. Είπατε ότι δεν είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε μαθήματα την πλευρά σας. Να σας πω κάτι. Οι πολίτες σας σας εξέλεξαν για να ακούσατε μαθήματα από την πλευρά μας. Όπως πρέπει να ακολουθήσω και μαθήματα από την δική σας πλευρά και τις ομιλίες σας. Και αυτό που δεν δέχομαι από εσά είναι ότι λέτε σε εμά εδώ ότι ξεχάσαμε τους θανάτους της 11 Σεπτεμβρίου. Ποτέ δεν θα σα πω ότι εσεί σκοτώνετε τι ελευθερίε, αλλά μην προσβάλλετε αυτή την πτέρυγα του Κοινοβουλίου λέγοντα ότι ρισμονήσαμε τα θύματα τη τρομοκρατία. Διακόπτη πρόεδρο, τον ε, ομιλητή. Δίνω το λόγο στην κυρία Βέρτμαν για ένα λεπτό. Όλοι πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ πρέπει να προστατεύουν την ασφάλεια όλων οι κοινέ διμερείς προσπάθειες δεν εξυπηρετούν. Συμφωνούμε όλοι. Πρέπει όμως να επαναλάβουμε ότι η συμφωνία των δεδομένων ρυθμίζεται στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα άρθρα 13 και 21 θα πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα στη συμφωνία αυτή γιατί ε, είναι σε αντίφαση το ένα προς το άλλο και δεν προσφέρουν νέα δικαιώματα στους πολίτες. Παρακαλώ την Κομισιόν να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή λύση. ελευθερία χωρίς ασφάλεια είναι εύθραυστη, κατασταλτική όμως είναι και η ασφάλεια χωρίς ελευθερία. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία και με την προσπάθεια όλων μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο κύριος Έγγελ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από αυτή τη συζήτηση τόση ώρα θεωρώ ότι δυστυχώ αυτή η συμφωνία δεν σχετίζεται τόσο πολύ με θέμα ιδιωτικότητα ή ασφαλεία, αλλά περισσότερο αφορά το να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για να μπορεί να ισχύσει η ανταλλαγή των δεδομένων. Είναι δυνατόν να κάνει ό,τι θέλουν, ε, είπα, Και επομένω, όποιο θέλει να πάει στην Αμερική θα πρέπει να αποφασίσει αν θα όχι με αυτό το πλαίσιο. Επίση, θα κάνουν ό,τι μπορούν οι Αμερικανοί για να αποσπάσουν ό,τι θέλουν. Και έχουμε επομένω μια τέτοια συμφωνία, η οποία τώρα ολοκληρώνεται. Δυστυχώ όμω δεν έχουν καμία συνθήκη Λισαβόνα, είπα, σε σχέση με την κύρωση συμφωνιών. Αυτή τη συμφωνία τη συνήψε ο πρόεδρος τον είπα. Επομένως δεν μπορεί να ρυθμίσει δικαιώματα τα οποία δεν προϋπάρχουν δυνάμει του Αμερικανικού δικαίου. Επομένως, δεν μπορώ εγώ να πω ναι μια συμφωνία η οποία δεν αλλάζει τόσα ισχύουν. Δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα, καμία διαφορά δεν θα έχει μεταχείριση των ε, επιβατών. Τίποτα δεν θα βελτιώσει ή δεν θα χειροτερέψει αυτή η συμφωνία. Ούτε πρόκειται να υπάρχει καμία καλύτερη προστασία δεδομένων από ό,τι ισχύει σήμερα, διότι εάν χρειαστεί, οι Αμερικανοί θα πούν ότι οι Ευρωπαίοι επιβάτες ε, θα πρέπει να με το Αμερικανικό Δίκαιο. Λυπάμαι, δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δρούτσα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να το πούμε ξεκάθαρα, η συμφωνία δεν είναι τέλεια και τα επιχείρηματα, ιδιαίτερα επιφυλάξει που εκφράστηκαν και σήμερα, σίγουρα έχουν βάση. Το θέμα όμω είναι το εξή. Ποια είναι η εναλλακτική λύση, με ποιον τρόπο κατοχυρώνουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπό τι παρούσε συνθήκε ε, βέβαια η απάντηση πιστεύω είναι με αυτήν την συμφωνία που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε με όλες τις αδυναμίες της τις οποίες γνωρίζουμε καλά. θα ήθελα όμως να αναλογιστούμε και ένα άλλο στοιχείο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο καλείται σήμερα να ψηφίσει μια διεθνή συμφωνία και σε μια διεθνή συμφωνία πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι όπως ποιο είναι το μέλλον ε, της συνεργασίας της ευρωπαϊκής ένωσης με τις ηπα ποιο θέλουμε να είναι ο ρόλο ε, τη ευρώπη στι διεθνεί εξελίξει στο μέλλον το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διεκδικεί ορθώ έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στι διαπραγματεύσει διεθνών συνθηκών τη ένωση και πρέπει ω ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να έχουμε αυτόν τον ρόλο στο μέλλον. πρέπει όμω να αποδείξουμε ω ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ότι είμαστε υπεύθυνοι και ξέρουμε και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι ευθύνε μα. ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δίας Δεμέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η, άποψή μου είναι η εξής. Όσον αφορά τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η συμφωνία PNR είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και τώρα αποτελεί ένα κομμάτι της στατικής Ευρωπαϊκής Ενώσης κατά της τρομοκρατίας, ε, αποτελεί ένα κομμάτι της στατικής Στοκχόλμης που μιλά για ανάγκη στενή συνεργασίας με τίτες χώρες συμπεριλαμβανομένης ανταλλαγής πληροφοριών. Στοιχεία θα συλλέγονται μέσω της συμφωνίας PNR και θα χρησιμοποιηθούν για πρόληψη, διερεύνηση, δίωξη τρομοκρατών, ε, εξυχνίαση σοβαρών εγκλημάτων είναι μια βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία του 2007. Η μέθοδος πού πρόθεση στοιχείων, αναγνωρίζεται σαν ένα πρότυπο, θα υπάρχει καλύτερη προστασία των συλλεγωμένων στοιχείων, θα έχει η εποπτική αρχή περισσότερες εξουσίες και θα υπάρχει και βελτίωση στην προστασία όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων. Οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα διορθώσεων και αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ε, διοικητικής ή δικαστική αποκατάσταση αποζημίωση θα είναι δυνατή η συμφωνία αναγνωρίζει τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτική ζωής, αναγνωρίζονται στην αρχή τη αναλογικότητα και αυτό ευθυγραμμίζεται με τους στόχους ε, των κοινών συμφερόντων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων. Μπορούμε να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία και να ωφεληθούμε από τις βελτιώσεις που επιφέρει ή να καταψηφίσουμε τη συμφωνία προξενώντας ένα νομικό κενό και θα δούμε διάδοση και αύξηση των διμερών συμφωνιών και θα δημιουργηθεί ένα νομικό κενό για τις αεροπορικές εταιρείες. Θα πρέπει να εργαστούμε για ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία των δεδομένων και δίποτε διαβίβαση στοιχείων PNR προς τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα εντός ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου, θα πρέπει να προστατεύονται δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω στοιχείων. Πρόεδρε, είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας για όλους αυτούς τους λόγους που εξασφαλίζει την καταπολέμηση του Εθνούς εγκλήματο και την τρομοκρατία. Δεχόσαστε από πλευρά του κύριου Λάιτφριντ ερώτημα σύμφωνα με τη διαδικασία τη γαλάζια κάρτα. Δεχόσαστε, ναι, κύριε Λάιτφριντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντίας Ντεμέρα, Μιλήσατε για τη στρατηγική της Ένωσης κατά της τρομοκρατίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμεθα. Όμως οι βασικές, οι θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών σε αυτό το πλαίσιο περιορίζονται συνεχώς. Έχουμε το SWIFT, έχουμε την ACTA, τη συμφωνία αυτή τώρα. Δεν ανησυχείτε ότι στο τέλος ε, θα ε, ε, ε, λειτουργήσω με κάθε υπερβολή με αυτόν τον τρόπο. Εγώ φοβάμαι όταν θα έρθει ε, μέρα που θα το διαπιστώσουμε αυτό. Ευχαριστώ αξιότιμε συνάδελφε. Πραγματικά αυτό που ήθελα να πω, ίσως δεν με ακούσετε προσεκτικά, αναφερόμουν στη στατική ασφαλεία Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Εσείς χρησιμοποιήσατε διαφορετική γλώσσα. Εγώ χρησιμοποιώ τη γλώσσα του Θερβάντες. Επικοινωνούμε μέσω διερμηνίας, αλλά δεν επικοινωνούμε λόγω διαφορετικών γλωσσών. Εσείς μιλούσατε για ιδεώδη, εγώ μιλούσα για εμπειρία που αντλώ από τον τομέα της ασφαλείας. Και βάσει τη δική μας εμπειρία στον τομέα της ασφαλείας, εγώ είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας. Για δύο λεπτά επόμενος ο η κυρία με Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω επί δύο πτυχών που θεωρώ σημαντικές δεν είμαστε εχθρικοί όσον αφορά το PNR εν γέννη και γενικότερα η καταπολέμηση τρομοκρατίας παραμένει μία από τις μέρημνέ μα τι σημαντικές, τι βασικές βάσει αυτών μπορούμε να πούμε ότι τελικά συμβιβασμό είναι και αυτό αποτέλεσμα παραχωρήσεων, άρα είναι ατελέ, αλλά δεν μπορεί να γίνει ει βάρο ενό μέρου από τα δύο συμβαλόμενα. Αυτή η εντύπωση κυριαρχεί και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να τα αρνηθούν. Σε αυτό το στάδιο τα επιχειρήματα που προβλήθησαν δεν πείθουν όλου να υπερψηφίσουν αυτή τη συμφωνία. Αν έχουν επιτευχθεί οι πρόοδοι, παραμένουν ανεπαρκεί και που δεν είδε καθησυχάζουν τι εκφραστήσει ανησυχίε που εκφράστηκαν ε, τον, Μάιο και τον Νοέμβριο του 2010 από το Κοινοβούλιο. Χρειάζεται αναλογικό πραγματικότητα. χρειά... δεν είναι σαφή η σκοπή, η διάρκεια κράτηση των στοιχείων, υπερβολική πεδία εφαρμογή πάρα πολύ ευρύ, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγή δικαστική, άρα μπορούμε να βάλουμε τα διάφορα μειονεκτήματα σε μακροσκελή κατάλογο. Αυτό είναι λυπηρό, διότι αυτή η συμφωνία θα έπρεπε ε, να οδηγήσει υψηλά επίπεδα προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια είναι η λογική τη δήλωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα μα υπόσχεται το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά, ε, ευτυχώ. Μα λένε ότι το Κοινοβούλιο ευδεί ελλείμματα στη συμφωνία και ζητεί αναστολή. Δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικότατα αυτό το αίτημα. Ευτυχώ. Θα ήταν παράδοξο επί μήνε να λέμε ότι είναι διαπραγματεύσιμη αυτή η συμφωνία και να μα λέει μετά τι μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι τελικά για αυτού του λόγου θα καταψηφίσω αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Κύριε Σκοέλιο, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Δεν διατηρώ καμία αμφιβολία. Δεν διατηρώ καμία αμφιβολία ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ ΕΕ όσον αφορά το PNR είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Καλύτερη από τι ε, διμερεί ε, συνθήκες. Και έτσι θα έχουμε περισσότερη συνέπεια, περισσότερη ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ε, συμπολιτών μας. Το τελικό αποτέλεσμα, Επίτροπε, όμως, απέχει πάρα πολύ από όσα θα θέλαμε και θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει. Κοιτάξτε τι ισχύει. Πρώτα πρώτα. Δεν έχουμε καμία καλύτερη προστασία από ότι πριν των δικαιωμάτων των, των, ε, των Ευρωπαίων. Μερικοί λένε ότι έτσι έχει βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η, ε, οι κανόνε κατακράτηση των δεδομένων και διάφορα άλλα σημεία. Όμω, εγώ σα παραμένω στο σημείο 21 τη συμφωνία που λέει ότι ε, ε, μπορεί να ε, που λέει τους όρους τέλος πάντων χρήσης αυτών των, των δεδομένων και έχουμε και το ζήτημα ε, του συστήματος πουλ, το ζήτημα της έγκρισης από το Κογκρέσο έχουμε και το σύστημα push που επίσης με, με την Αυστραλία εδώ όμως είναι το πουλ επομένως πρόκειται για κάποιο κυρίαρχο κράτος όπως είπα έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για το ποιος εισέλθει στην επικράτειά τους όμως το ζήτημα είναι ε, το, το αν ε, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους ε, συλλογή στοιχείων από τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μας. Είναι ευαίσθητα αυτά τα δεδομένα. Έχουμε τη συμφωνία του 2004 που απειγόρευε τη χρήση αυτών των δεδομένων. Τώρα όμως επιτρέπεται η κατακράτηση δε αυτών των δεδομένων τώρα έχει παραταθεί. Πάμε προς αόριστη περίοδο κατακράτησης. Ευχαριστούμε τους ηγητές Ευχαριστώ πολύ, λέει σας όλοι. Επίτροπε Μάστρομ, καλά το είπατε. Δεν είναι τέλεια συμφωνία. Αν δεν είχαμε κάνει εμείς οι Ευρωπαίοι, θα είχαμε ακολουθήσει διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτή δεν είναι μια οδηγία, είναι μια συμφωνία, συμφωνία μεταξύ μερών. Συμφωνία είναι πάντα καλύτερη από μη συμφωνία και είναι μια συμφωνία αυτή που μας οδηγεί σε βήματα πρόοδου. Βήματα πρόοδου που μπορούν να επιτρέψουν και μεταγενέστερες βελτιώσεις, διότι κάθε χρόνο χωρίς μυστικές συμφωνίες όπως έχουν γίνει με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία θα επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και θα επαληθευτεί, θα ελεγχθεί στο Κοινοβούλιο. Είναι ένα πολιτικό στοιχείο αυτό. Η Ευρώπη με αυτή τη συμφωνία είναι στο τραπέζι συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ και μπαίνει στην Αμερικανική νομολογία. Ευχαριστώ την ομάδα μου που επέτρεψε ελεύθερη ψήφο και την αντιπροσωπεία του δημοκρατικού, Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος ε, που θα υπερψηφίσει την ε, συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Σασόλη. Πάμε στη διαδικασία απόσπαση προσοχή της Προέδρου. Α, γαλάζια κάρτα. Α, για το ΚΑΣΤΙΑ, για το απόσπαση προσοχή. Δεν μπορώ να ε, δεχτώ όλο τον κόσμο γιατί έχουμε και άλλη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε την κυρία Κοράτζα. Παρακαλώ τηρήστε το χρόνο στη διάθεσή σα. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Εκτό μικροφώνου κύριε Κόρατσα. Μικρό, μικρό. Vous me faites recommencer. Oh, voilà, merci. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και δεν άκουσα όμως με μέσα σε όλη αυτή την κριτική μία ρεαλιστική εναλλακτική. Τι γίνεται με τις διεθνείς δεν ξέρετε. Πρόκειται περί συμβιβασμών. Είναι σαν σαν το χορό. Ο ένας με τον άλλο. Και εσείς τι αναλεκτή έχετε να προτείνετε. Τι να κάνουν οι Ευρωπαίοι, να μην ταξιδεύουν στη ΣΥΠΑ. Να, αυτό τους λέτε ουσιαστικά. Αυτό όμως είναι αποστέρηση ελευθερίας. Επομένως, ε, ας είμαστε πια λίγο, λιγουλάκι ρεαλιστές. Δεν είναι ιδιώδης αυτή η συμφωνία. Σύμφωνη. Τι άλλο όμως υπάρχει. Οι ΗΠΑ μπορούν να συλλέξουν δεδομένα στη χώρα τους. Στη χώρα τους πάνε να ταξιδέψουμε. Τι προτιμάτε, μυστικές διμερείς συμφωνίες με κράτη-μέλη. Θέλετε να μη δίνουν θεωρήσεις διαβατηρίων. Αυτό θα γίνει. Έχουμε βελτίωση σχέση με το 2007. Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Εγώ είμαι υπέρ. Διότι τώρα έχουμε εγγυήσει, έχουμε ασφάλεια για του Ευρωπαίου. Ευχαριστώ. Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συμφωνία πάσχει σε σημαντικά σημεία. Οι Ευρωπαίοι τώρα αποστερούνται του δικαιώματος προσφυγής στα Αμερικανικά δικαστήρια. Όμω την καλύτερη αυτή συμφωνία από την προηγουμένη και καλύτερη από τι διμερεί συμφωνίε. Για μα, του Πορτογάλου, η κυβέρνησή μα έχει κυρώσει μια συμφωνία. Αλλά εκείνη η συμφωνία ήταν πολύ χειρότερη τη παρούση. Εάν το Κοινοβούλιο δεν δώσει το πράσινο φω, θα έχουμε ένα σωρό χειρότερε, πιο περιοριστικέ συμφωνίε. Εάν πούμε ναι, θα έχουμε περισσότερη προστασία των Ευρωπαίων. Και έτσι μπορούμε να ε, συμπράξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την συμφωνία. Ο επόμενος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, και Κύριο κύριος είμαστε αποφασισμένοι πιο αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και μέσα πρέπει να λάβουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία όμως να συνάδουν προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να μην έχουμε χρήση και κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων. Θα πρέπει επίσης να σεβαστούμε την αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, η συλλογή, η επεξεργασία και κατακράτηση των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνεται επί τη βάση κάποιων αυστηρών κανόνων. Θα πρέπει επίσης να διέπεται από κάποια εποπτεία και έλεγχο. Πολλά ακόμα είναι σκοτεινά σε αυτή τη συμφωνία, γι' αυτό και νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε τις εγγύσεις που θέλαμε. Πάσκου. Η σημερινή συμφωνία εκφράζει μια νέα ισορροπία μεταξύ ενός κράτους που θέλει όλο και περισσότερο ερευνά ε, και περιορίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Δεν θα πω στις τεχνικές λεπτομέρειες. Τρία να πω. Πρώτον, πριν ασχοληθούμε με τη μεταφορά των στοιχείων PNR, έπρεπε να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο τους κατά τη συλλογή τους. Δεν βλέπω τι σχέση έχει όταν κλείνω ένα εισιτήριο, ε, το αν συμμετέχω σε ένα συνδικάτο. Συλλέγονται στοιχεία στην Ευρώπη. Δεν μεταφέρονται μονομένα. Θέλουν οι Αμερικανοί τα στοιχεία να τα συγκρίνουν τα δικά του. Που ήδη έχουν συλλεχθεί με άλλου τρόπου. Λαμβάνοντα αυτά υπόψη, φοβούμαι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Παρά να εγκρίνουμε όμω τη συμφωνία και αυτό που να κάνουμε. Ο κύριο Σαλβάρμα έχει το λόγο. Σε 9 το πρωί κάθομαι εδώ πέρα. Και έχω μείνει έκθαμβος. Δεν άκουσα δύο πράγματα. Εφαρμογή του νόμου. Δύο λέξεις. Πήγαμε πιο ένα καφεδάκι πριν μερικά λεπτά. Ίσως όταν έλειπα να αναφέρθηκε αυτό. Όπως και ο κύριος Κέρκοπ είπε με τα έξοχα σχόλια του, δεν είναι Αμερικανός, ούτε εγώ είμαι Αμερικανός, αλλά έχω ζήσει στη ΣΥΠΑ αρκετά χρόνια. Και φοβούμαι ότι κάποια στοιχεία της σημερινής συζήτησης αντικατοπτρίζουν σοβαρή παρεξήγηση κινητών και προθέσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιους από τους αγορητές στην αριστερή πτέρυγα του ημικυκλίου. Αν έρθει κάποιο σπίτι σας, δεν σας ενδιαφέρει ποιοι είναι, τι θέλουν εκεί. Δεν σας ενδιαφέρει ποια είναι η πρόθεσή τους, ποιο είναι το κινητρό τους. Είναι παράλογο νομίζω. Εγώ θα ενδιαφερόμουν. Δεν καταλαβαίνω το όλο θέμα. Εγώ θα υπερψηφίσω. Είναι σαφέ. Ευχαριστώ, κυρία Μέσνερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πολύ σέβομαι τις προσπάθειές σας για βελτίωση της συμφωνίας που έχει τη μορφή την τωρινή, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα μπορούσα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο προλαλής σας. Βεβαίως ε, θέλουμε να ξέρουμε τι θέλει ένας άνθρωπος που έρχεται στο σπίτι μας, αλλά τα στοιχεία του δεν τα κρατάμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είπατε μετά από έξι μήνες γίνονται ανώνυμα. Εντάξει, αλλά επί έξι μήνες δεν είναι. Πολλά, πολλές επιφυλάξεις πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είπατε ότι τα δεδομένα συλλέγονται ούτως ή άλλως. Αυτό δεν είναι λόγος για μένα για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να βιαστούμε και με τις διαπραγματεύσεις, με τις υπά, Βεβαίως πολλά δεν είναι ε, ισορροπημένα και σωστά όπως τα στοιχεία που συλλέγουν και μεταδιαβιβάζουν διαβιβάζουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ίσως ε, είναι καλύτερα να μην έχουμε συμφωνία παρά να έχουμε κακή συμφωνία. Η κυρία Πρέντεργκαστ. Συνάδελφοι, έχω πάρα πολύ σοβαρέ επιφυλάξει σε σχέση με τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά το, το, αν χρειάζεται για τις μεθόδους για το, για το, για το της και είπαμε ότι δεν έχει αποδειχθεί με τίποτα η αναλογικότητα και για το ότι τι θα γίνει η ε, πρώτη περιγύρωση χώρα και επομένω ζητάτε τι απαραίτητε πληροφορίε για αυτού που θα μπουν στην επικρατεία τη. Εγώ έχω θεωρήσει ότι η Επίτροπος όμως ε, ε, διαπραγματεύτηκε ό,τι μπορούσε για εγγυήσεις για τους πολίτες της Ευρώπης. Και αν ε, απορρίψουν τη συμφωνία δεν θα σταματήσουμε τη είπα, να έχουν πρόσβαση στις τις πληροφορίες στα δεδομένα μας και αν δεν θα έχουμε καμία εγγύηση. Άρα θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Ε, αν θέλουμε εμείς να είμαστε υπεύθυνοι και λογικοί. Ευχαριστώ. Μπένοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, τα είπαμε σχεδόν όλα. Και θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο εάν τελικά αυτή η ζήτηση εξελισσόταν σε συζήτηση μεταξύ Αμερικανών και αντιαμερικανών, ε, φιλοαμερικανών και αντιαμερικανών. Και επομένω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι βελτιώνεται η αρχική συμφωνία. Είχαμε πει όχι το Μάιο. Και δηλαδή, μεριά να λάβουμε υπόψη το ότι η, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ τρομοκρατία και έγκλημα, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη συνεργασία. θα μπορούσατε να πετύχετε περισσότερα, κυρία Επίτροπε. Έχει πολλά δυνατά σημεία αυτή η συμφωνία. Δεν μπορώ να την ψηφίσω. Κυρία Λάτφορντ, θα ήθελα η κυρία Επίτροπος Μάλστρεμ ότι εκτιμά τα μάλα η Άλντε το έργο της. Και επίσης σημαντικό κομμάτι της Άλντε να υπερψηφίσει τη συμφωνία. Αυτό. Και η δήλωση που μας προσέφερε ε, είναι πολύτιμη. Πιο συγκεκριμένα, οι υποσχέσεις παραναθεωρήσεως και μηχανισμού ελέγχου που θα συμπεριβάλλονται στη συμφωνία. Κυρίως πεδίο εφαρμογής και περιορισμός του δυνάμει το Άρθρο 4, διότι γνωρίζει, όπως και το Κοινοβούλιο, για τα 4, 2, 3 και 4 Και πιστεύω θα επαγρυπνεί για αυτά. Και όπως υποσχέθηκε θα επανέλθει σε εμάς για το θέμα αυτό. Στην πρώτη αναθεώρηση και στις επακόλουθες. Εκτιμώ τα όσα έκανε. Με έπεισε και άλλους να υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Λάτφορντ. Ο κ. Πάσκα έχει το λόγο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ συνήψαν συμφωνία για τη χρήση και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων για να νομιμοποιήσουν την επεξεργασία των ε, προσωπικών δεδομένων των ε, Ευρωπαίων πολιτών από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ. Ε, τον περασμένο Μάιο αρνηθήκαμε να εγκρίνουμε τη συμφωνία γιατί δεν λαμβάνονταν υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ρυθμίζουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το νέο κείμενο της συμφωνίας που συζητάμε σήμερα βελτίωσε την ε, προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία τους με νομότυπο τρόπο. Το νέο κείμενο παρόλα αυτά έχει ελλείψεις που ήταν ο λόγος που απορρίφθηκε τον περασμένο Μάιο. Τώρα θα πρέπει να ε, το θεωρήσουμε προσπάθεια επίτευξης ε, ε, συμβιβαστικής λύσης. Πιστεύω, κυρία Επίτροπε, όμως ότι δεν έχουμε πλήρη προστασία όπως θα έπρεπε. Κάτι διαδικαστικό, συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά μου λέγουν ότι γερμανική και η αγγλική μετάφραση έκανε ένα λάθος στην παρέμβασή μου. Είπα ότι δεν μπορώ να εγκρίνω αυτή τη συμφωνία και εξήγησα τους λόγους. Αλλά αναφέρθηκε διαφορετικά, μεταφράστηκε αντιθέτως αυτό που είπα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι θα απόσχω, όπως είπα και στην παρέμβασή μου. Ευχαριστώ, σημειώνουμε δεόντως Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη. Πού είναι τα όρια όσον αφορά αυτά που μπορούμε να ανεχθούμε και αυτά που μπορούμε να επιτρέψουμε στη ΣΥΠΑ να μας επιβάλλει να μας επιβάλλει τις προδιαγραφές τους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την ε, προσπάθεια καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και της Πέρασαν κάποιους ε, όρους ε, που δεν έχουν σχέση με την καταπολέμηση της Επί δέκα χρόνια τελούν υποκράτηση στη ΣΥΠΑ άνθρωποι χωρίς να δικαστούν. Και αυτή η πρακτική είναι απαράδεκτη για μας δεχτήκαμε παρόλα αυτά να κατασκευάσουν μυστικές φυλακές και να συνεχίσουν αυτή την πρακτική εκεί. Ίσως η συζήτηση δεν είναι πολύ σχετική στον αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων το λέω για να, να τραβήξουμε τη γραμμή. Η συγγήτρια, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μιλήσουν και μετά έχουμε και συζήτηση πριν ψηφοφορία. Πρέπει να προχωρήσουμε, συγγνώμη. Διαδικαστικό, ρωτάει ο Πρόεδρος, ο κ. Γκότφριντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν αμφισβητώ τον τρόπο που προεδρεύεται, που είναι εξαιρετικός, μία πρόταση ίσως για το μέλλον και εγώ ζήτησα το λόγο για, στη διαδικασία Catch the Eye ε, από την αρχή μάλιστα. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να δίνετε στο το, λόγο σε όσους παρακολούθησαν όλη τη συζήτηση και όχι σε όσους ήρθαν την τελευταία στιγμή. Το σημειώνω, δύσκολη ημέρα. Έχω και χρόνο διάγραμμα να τηρήσω. Έχουμε ψηφοφορία στι 12 και έχουμε μετά το εμπόριο Λευκής Αρκός, το εμπόριο ανθρώπων να συζητήσουμε. Ζητώ συγγνώμη. Δίνω το λόγο στην κυρία Μάστρομ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλου. Πολύ καλή συζήτηση. Άριστη συνεργασία με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών ε, και τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον, δυο Πεδίο εφαρμογή τώρα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα ε, που οδηγεί σε ποινές τρία χρόνια. Δεν έχουμε μετανάστευση, μεθοριακό έλεγχο κλπ. σαν πρόσθετου στόχου. Προστασία ζωτικών συμφερόντων όσον αφορά θέματα ζωή ή θανάτου, μεταδοτικέ ασθένειε, Αυτά συνέβησαν σε τέσσερι περιπτώσει μόνο κατά τη διάρκεια τη αναθεώρηση που κάναμε στην ισχύουσα συμφωνία από το 2007 μέχρι το 2010. Σε τέσσερι περιπτώσει και καμία αυτέ τι περιπτώσει ενέπλεκε στοιχεία PNR. Όσον αφορά δικαστικά εντάλματα, στο Σύνταγμα των ΗΠΑ και σε κάποια από τα ευρωπαϊκά συντάγματα, ένα δικαστήριο μπορεί να ζητήσει στοιχεία PNR να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί ότι κάποιο ήταν σε ένα αεροπλάνο ή όχι. Μόνο μια φορά αυτό συνέβη Αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες ε, και όλες έχουν καταγορηθεί και καταγραφεί. Όσον αφορά το push και το pull, άντιση και αποστολή πληροφοριών. Το πρότυπο είναι η αποστολή, το PUS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροπορικών ε, Εταιριών και Διεθνέο Οργανισμό το δέχτηκαν, το θεώρησαν ευπρόσδεκτο και τεράστια πλειοψηφία των αεροπορικών εταιριών χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο και θα μπορούν να συμμορφωθούν και με την απέτηση να έχουν τη δυνατότητα πρόθεση πληροφοριών εντό διετίας. Όσον αφορά την αποζημίωση αποκατάσταση, αναφέρθηκε ότι στη συμφωνία ότι οποιοδήποτε μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο κατά αποφάσεω που αρνείται πρόσβαση λόγω στοιχείων ε, βάσει της, του νόμου για την ελευθερία των πληροφοριών. Η ονομοθεσία στη ΣΥΠΑ δεν είναι αυτό το δικαίωμα στους Αμερικανούς. Αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα για αποφάσεις που λαμβάνει η Αμερικανική κυβέρνηση και μπορεί να αναθεωρηθεί δικαστικά ε, να εξεταστεί δικαστικά και να δοθεί αποζημίωση για το περιεχόμενο των στοιχείων. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι αυτά που δίνεται όταν κλείνεται μια αεροπορικό εισιτήριο. Ε, δεν αναφέρεται εκεί αν είσαστε μέλος συνδικάτου ή τι θα ψωνίσετε στο αεροδρόμιο. Αυτά τα στοιχεία που δίνεται καταχωρούνται. Δεν ξέρω πόσο ενήμεροι είναι οι επιβάτες περί αυτού, αλλά λέμε στη συμφωνία ότι είπα πρέπει να πληροφορούν τους επιβάτες περί αυτού. Αυτή είναι η σοβαρή βελτίωση. Όσον αφορά την εικόνα του, το, για το άτομο, για τη στοιχεία του ατόμου, σχηματισμό εικόνας αυτά απαγορεύονται. Οι ΙΠΑ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν στοιχεία από ένα άτομο που θέλει να μπει στη χώρα τους. Το κάνουν σήμερα, το έκαναν κατά το παρελθόν και θα το κάνουν και στο μέλλον. Όπως το κάνουν και τα περισσότερα κράτη-μέλη. Και διαπραγματευόμαστε τώρα και το συζητήσουμε αργότερα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως PNR, γιατί τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό είναι πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά πιο σημαντικό λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ανθρώπων. Καταπολεμούνται με αυτόν τον τρόπο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλουμε η μεταφορά των στοιχείων να χρησιμοποιείται αναλογικά, περιορισμένα, με τη μέγιστη δυνατή προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ακεραιότητα ατόμων. Αυτή είναι η άποψή μα Ζητήσατε αδιαπραγμάτευση τη συμφωνία του 2007 που ισχύει σήμερα. Το κάναμε. Όλοι μαζί. Με τη στεναρή σα υποστήριξη. Με σαφείς κατευθύνσεις. Μέσω του ψηφίσματό σας και με την υποστήριξη του Συμβουλίου. Δεν είναι τέλεια συμφωνία. Όχι, δεν πήρατε 100% αυτά που ζητήσατε. Όμως, σε όλα τα σημεία είναι καλύτερη η συμφωνία από την ισχύουσα. Και γι' αυτό ζητούμε να την υποστηρίξετε, να την ψηφίσετε. Προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτή τη συμφωνία, όπω όλοι σα. Θα την αναθεωρήσουμε και στην αναθεώρηση, κύριε Σίγκμπερ, θα υπάρχουν εμπειρογνώμονε για την προστασία των δεδομένων παρόντε. Και δεσμεύομαι, όπω και στην πρώτη έρευνη δήλωση, ότι θα επικρατήσει πλήρη διαφάνεια και θα σε ενημερώνω ε, σε όλα τα βήματα που θα ακολουθούμε όσον αφορά τι αναθεωρήσει. Ευχαριστώ, κύριε Μάστρο. Με του, του Συμβουλίου, ο κύριο Μπότσκοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και πάλι πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετέχω στη συζήτηση. Είναι σημαντικό το θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης και είδαμε πάλι ότι όλοι θεωρούμε το ζήτημα αυτό σημαντικότατο. Όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το θέμα δεν είναι απλό και πολλές ανησυχίες που εκφράστηκαν συζητήθηκαν ε, με μεγάλες λεπτομέρειες. Όπως και η Επίτροπος Μάλμστρομ, θα ήθελα και εγώ να θεωρήσω ε, δεδομένο ότι η Προεδρία θεωρεί ότι η συμφωνία είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Αν αποτελεί βελτίωση η τωρινή συμφωνία σε σχέση με την προηγούμενη, δηλαδή αν θα έχουμε ευκαιρίες να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας να καταπολεμήσουμε τη το διασυνοριακό σοβαρό έγκλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι πολύ εξημών έχετε επιφυλάξεις επί του σχεδίου συμφωνίας αλλά ελπίζω ότι και εγώ και η Επίτροπος Μάλμστρομ ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα. Βεβαίως θα εξετάσουμε και τις επιφυλάξεις και όλες τις ερωτήσεις σας με πολύ ε, σοβαρότητα, αλλά πολλές απόψεις που ακούσαμε σήμερα συζητήθηκαν βέβαια και στο Συμβούλιο. Αλλά και πάλι συμπερασματικά επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι το τέλος του διατλαντικού διαλόγου για τη χρήση των πληροφοριών PNR. Έχουμε συμφωνία για την αξιολόγηση και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ευκαιρία να δούμε αν οι διατάξεις της συμφωνίας τηρούνται στην πράξη και όταν πρόκειται και για περιορισμούς χρήσης. Οπότε πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση για τα, η χρήση των PNR μπορούμε να έχουμε βελτιώσεις και θα αντιμετωπίσουμε και ένα κατεπήγον πρόβλημα που ε, ε, αφορά τους πολίτες και τις αεροπορικές εταιρείες. Όπως είπε η Επίτροπος Μάλμστρομ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμμετέχουν και θα ενημερώνονται ε, όταν αξιολογήσουμε την ε, συμφωνία και ε, βεβαίως για λογαριασμό του Συμβουλίου συμφωνώ με αυτό. Ευχαριστώ που επιτρέψατε να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση και ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Και τώρα η συγγήτρια, η κυρία Ιντφέλτε. Πολύ σύντομα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διαλύσω μια παρεξήγηση που την έχω επαναλάβει χιλιάδες φορές. Κανείς δεν αμφισβητεί εδώ την ανάγκη να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού ε, διασυνοριακού εγκλήματος, κυρία Φώστερ. Αλλά δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται για άλλα, όπως μεταδοτικά νοσήματα και ελέγχου ε, από το τμήμα μετανάστευσης και τα τελωνία. Εσείς έχετε κάποια ερμηνεία για το άρθρο 4. Η ερμηνεία αυτή όμως δεν είναι ίδια ε, για όλους και θα ήθελα ε, να ξέρω εάν τη συμμερίζονται ή είπα και πώς το ξέρουμε αυτό. Επίσης προς την κυρία Κοράτσα Μπίλτε, βεβαίως ε, ε, οι διεθνείς συμφωνίες σημαίνουν συμβιβαστικέ λύσεις, αλλά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κοινωνικό δίκαιο δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Ε, γιατί με την Αυστραλία έχουμε ε, καταφέρει να έχουμε καλή συμφωνία με τους Αμερικανούς συμμάχους και τους εταίρους όχι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Η ανάλυση του κυρίου Έγγελ από το ΕΛΚ ε, είναι ότι χωρίς τη συμφωνία θα έχουμε λιγότερες εγγύησεις ε, όμως ακόμα και αν καταψηφίσουμε τη συμφωνία έχουμε ε, ε διασφαλίσεις και εγγύσεις. Για το push και pull ε, δεν είναι όλες οι εταιρείε πρόθυμες να περάσουν στο push και ξέρουμε ότι αυτή η ρήτρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ακόμα και αν ισχύει η μέθοδος push όπως ισχύει ε, όπως προβλέπετε, εξακολουθεί να υφίσταται και η μέθοδος πουλ και οι Αμερικανοί θα πάνε στους κομπιούτερ και θα πάρουν τα δεδομένα. Δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου γιατί ε, ε, τι, γιατί λέτε ότι είναι ε, εξαίρεση οι χιλιάδες μέθοδοι πουλ που χρησιμοποιούνται κάθε μέρα. Γιατί λέτε ότι είναι κατεξαίρεση. Τέλος για την παρακολούθηση. Αν η εμπειρία από τη συμφωνία SWIFT και η παρακολούθησή της έχει κάποιο νόημα, η παρακολούθηση είναι ένα αστείο, είναι αστεία. Τέλος, αναρωτηθείτε. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και ρωτήστε αν άλλε χώρε χτυπήσουν την πόρτα μα και ξέρουν ότι θα το κάνουν. Το Κατάρ το έκανε. Η Ιαπωνία επίση, η Νότια Κορέα, η Κούβα θα ακολουθήσει, η Νότια Αφρική θα ακολουθήσει, η Κίνα, η Ρωσία επίση, Είμαστε διατεθειμένοι να τους δίνουμε τα δεδομένα τους και να τα χρησιμοποιούν για profiling με τους ίδιους όρους όπως κάνουμε τώρα για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό είναι ερώτημα κέριο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε στις 12 Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μέτσας Διατάξεως, λέει ο Πρόεδρος, το οποίο αφορά τις δηλώσεις ε, Συμβουλίου και Επιτροπής σε σχέση με την ε, μεταχείριση των φυσικών προσώπων. Έχετε τον λόγο κύριε